Προτείνω να αρχίσουμε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν σχόλια, ανακοινώσεις. Να σας πω ότι εγκρίναμε δύο κατεπήγοντα για την κατάσταση στη Γουινέα Κονακρή ε, κατά των ε, διαδηλωτών και την ε, παιδική εργασία στη Μαδαγασκάρη. Όπως ξέρετε επίσης ε, ε, λάβαμε γνώση της απελευθέρωσης του νικητή του βραβείου Ζαχάροφ 2017, τον Λορέν Σαλέχα, τον οποίο θα δεχτούμε κιόλα και θα μας μιλήσει για την κατάσταση στη χώρα του και, το λεγόμενο λευκά, και τα λεγόμενα λευκά βασανιστήρια. Ο Λορέντ έχει ε, προβάλλει μία θεατρική παράσταση, την οποία και θα δούμε αύριο στις 18 Φεβρουαρίου στις 6.30. Θα ήθελα να συμμετάσχετε σε αυτή την συνάντηση θεατρική παράσταση. Επίσης, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ε, που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση για την κατάσταση στα σύνορα Αμερικής Μεξικού ότι η συνεδρίαση θα γίνει αύριο στις 5 ε, και 4, 5 και 4 με 6 και 4. Επίσης να υποδεχτούμε τον κύριο Κριστιαν Σαργάτς, νέο μέλος από το ΕΛΚ, από την Αυστρία, ο οποίος δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Τρία, Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 23ης Δεκεμβρίου, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Περνάμε στο σημείο 4. Τώρα έχουμε την παρουσίαση της κατάστασης για την βιοπικιλότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα και τις επιπτώσεις της στην εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε το θέμα έχει περάσει στο προσκήνιο των παγκοσμίων δρόμενων κατά το Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΜΚΟ πέρσι το Δεκέμβριο ασχοληθήκαμε με το ζήτημα και αυτό αφορά και την Σύμβαση για την Βιοπικιλότητα, η οποία θα συνεδριάσει τον Οκτώβριο 2020 και θα ασχοληθεί με θέματα βιοπικιλότητας μετά το 2020. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τη βιοπικιλότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα και τις επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρσι η Επιτροπή μας ζήτησε μία μελέτη που θα μας μιλήσει για το πολυσχηδές νομικό πλαίσιο με βάση τους στόχους και το ρυθμιστικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Θα δούμε λοιπόν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προβάλλει μία νέα προσέγγιση παγκόσμιας εμβέλειας Ως προς το θέμα αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μοργέρα, η οποία είναι καθηγήτρια στη Γλασκόβη και ε, είναι διδάκτορ ασχολούμενη με θέματα βιοπικιλότητας σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και την βιοπικιλότητα. Έχετε το λόγο και μετά εάν θέλουν να λάβουν το λόγο μέλη θα τον έχουν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντοπίζει αυτήν την περιοχή ως ε, ανάγκη προσπάθειας και καθορισμού προτεραιοτήτων. Στο 4,1 σημείο της μελέτης έχουμε όλο και περισσότερες αποδείξεις για τις ε, Πολλέ διασυνδέσεις μεταξύ των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιοποικιλότητα. και νομίζω προχωρούμε πολύ πιο πέρα του σκεπτικού της προστασίας του οικοστήματος ή της φύσης αλλά η προστασία της φύσης ενέχει τις δικές της επιπτώσεις κοινωνικές και πολιτιστικές πάρα πολύ διαδεδομένες και πολύ συχνά άμεσα συνδεδεμένες ε, με τους πιο ευάλωτους εξημών. Επομένως δεν πρέπει να βλέπουμε την προστασία της φύσης ε, ως αντίθετη προς τις ε, συνήθειες ή τα ήθη των κοινωνιών, αλλά ακριβώς ως πλαίσιο υποστήριξης τους και προστασία συγκεκριμένων πληθυσμών και συγκεκριμένων περιοχών. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικές αποδείξεις για το ότι είναι δικαίωμα όλων η υγεία. Αυτό είναι όλο και πιο κεντρικό σημείο σε διεθνείς συζητήσεις. Αυτό έχει μακρόπνοες επιπτώσεις, οι οποίες έχουν ε, μελετηθεί αρκετά και για πληθυσμού ηθαγενεί και για άλλους τοπικούς πληθυσμού που έχουν άμεση όμω σχέση με το οικοσύστημα, με τη φύση και που από τη φύση εξαρτάται το πολιτιστικό τους, πολιτισμικό του σύστημα. Επομένως είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή και είναι πολύ σημαντικό να επιτύχει. Επίσης έχουμε περισσότερη νομική σαφήνεια σαφήνεια δικαίου σχετικά με τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αλλά και της διεθνούς κοινότητας, πώς συνδέονται και σχετίζονται με νομικά δεσμευτικές διατάξεις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε πολλές και διάφορες δεσμεύσεις και διεθνείς υποχρεώσεις. Όλα αυτά έχουν στρατηγικό αντίκτυπο η κατανόηση του πώς η προστασία της φύσεως είναι θέμα του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιορίζει το περιθώριο ελιγμών νομικώς μιλώντας που θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα υπό τη σύμβαση της ε, βιοπικιλότητας που όλα τα κράτη-μέλη έχουν συνυπογράψει έχουμε αναπτύξει μια δέσμη βελτίστων πρακτικών από όλα τα συμμετέχοντα κράτη, περί τα 160, όπως και σχετικά με τις τοπικές και ηθαγενείς κοινότητες, αυτό είναι μια υγιής νομική βάση ώστε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση δράση επί του συσχετισμού μεταξύ της φύσεως και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και σε σημεία που θεωρούσαμε ότι είναι πιο απομακρυσμένα. Για παράδειγμα, προσέχουμε όλο και περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κλιματική αλλαγή, στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και έχουμε και καθοδήγηση για μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον άνθρωπο για την αντιστάθμιση της κλιματικής αλλαγής και για την προσαρμογή μας σε αυτήν. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί, έχουν συμφωνηθεί και παρέχουν πρακτικές συμβουλές και ασφάλεια δικαίου σχετικά με το πώς μπορούν να συντονιστούν διάφορες πηγές του διεθνούς δικαίου. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη μια βάση συνενετική για μια ολιστική προσέγγιση, λέει η ομιλήτρια, προς τους στόχους μας. η τροφή, το νερό, τα βασικά δικαιώματα των γυναικών, των ανηλίκων, των παιδιών και των ηθαγενών και τοπικών πληθυσμών είναι συστατικά του πλαισίου αυτού. Επίσης έχουμε ένα πλαίσιο καθοδήγησης για τις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της προστασίας της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των πόρων όπως και στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, της ε, χρηματοδότησης της έρευνας, της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας. Επομένως μπορεί κανείς να αντλήσει από όλα αυτά, από όλες αυτές τις δεξαμενές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από κοινού, από τα μέλη της διεθνούς κοινότητας και τα κράτη και μη κρατική φορείς. Η έκθεση λοιπόν εντοπίζει μια σειρά από ευκαιρίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για άλλους ε, φορείς και οργανισμούς ώστε να αναλάβουν δράση. Αυτό μπορεί να γίνει ε, δείχνοντας μια ηγετική θέση, δίνοντας το παράδειγμα θα λέει κανείς, στα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες. Γιατί ο συσχετισμός της φύσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημαίνει αρκετά περίπλοκες σχέσεις ισορροπίας. Χρειάζεται μια θετική προσέγγιση. Δεν είναι απολύτως εύληπτες σχέσεις αυτές για τα αναπτυσσόμενα κράτη. Έχω λοιπόν διακρίνει κάποιες συστάσεις πρώτον ε, ως προς το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή φόρα και υπάρχουν πάρα πολλέ ευκαιρίες σε συνεχιζόμενες διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Έθνη για να διερευνήσουμε την έννοια του πώς μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα η σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την βιοπικιλότητα βιοπικιλότητα στην οποία ε, διαπραγματευόμαστε ένα διεθνές πλαίσιο ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην προστασία της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης της, αλλά και άλλες διαδικασίες εντός της σύμβασης που μπορούν να υποστηρίξουν για τους ηθαγενούς πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες υπάρχουν πλαίσια συνεργασίας για τους ωκεανούς, για την κλιματική αλλαγή, όπου και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει σαφέστερο, εμφανέστερο ρόλο. Υπό τη Συμφωνία του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες για τις δασικές εκτάσεις ως προς την προσαρμογή, για τη χρηματοδότηση, για το κλίμα, για υποβολές προτάσεων που να βασίζονται στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα, λέει ο Μιλήτρια. Είναι εξίσου σημαντικό να δει κανείς ε, την βιοπικιλότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα στα χημικά απόβλητα, μεταξύ άλλων, έχουμε πολύ ακριβέστερη εικόνα για τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στη βιοπικιλότητα. Και συνεχίζονται οι συζητήσεις ε, στον ΟΗΕ για μια θαλάσσια σύμβαση ε, του δικαίου της θάλασσας. Οι ωκεανοί είναι απολύτως απαραίτητη για τους ε, στόχους βιωσίμου ανάπτυξης. Ωστόσο, πολύ σπάνια ακούμε κάποια, χάρη, κάποια χώρα με συγχωρείτε, να σημειώνει πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα με όλες τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια διεθνούς χρηματοδότησης έχει πολλές περισσότερες ευκαιρίες να οργανώσει την προστασία αυτή, τις διάφορες αυτές διεθνείς διαδικασίες ώστε να μπορούμε να δούμε τις ε, νομικές επιπτώσεις των διατάξεων αυτών, αλλά και για να υποστηρίξουμε μονομερείς και πολυμερείς ε, πρωτοβουλίες, ώστε να έχουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση, τροφοδοτώντας τα όσα μπορούμε να κάνουμε στο εθνικό επίπεδο προς το διεθνές και για να έχουμε διδάγματα για καλύτερες σχέσεις και πιο αποτελεσματικές με τρίτες χώρες. Οι συστάσεις επί των διμερών σχέσεων διαιρούνται σε δύο τμήματα. Είχαμε πολλή έρευνα για τα κεφάλαια εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης επί τη βάση των διμερών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί έχουμε ευκαιρίες για να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα στο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό δεν έχει ακόμα εγγραφεί, αν θέλετε, ως στοιχείο σε αυτές τις διμερείς συμφωνίες, αλλά υπάρχει περιθώριο στις διατάξεις υλοποίηση ώστε να δούμε τις αρνητικές επιπτώσεις και ώστε να υποστηριχθεί αυτός ο διάλογος και με ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την προστασία, την ωφέλεια που μπορεί να απορρέει από την προστασία της βιοποικιλότητας. Στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών, η χρηματοδότηση που σχετίζεται με την πλήρη του υλοποίηση και οι συμμετοχικές διαδικασίες που ξεκινούν υπό τις συμφωνίες αυτές είναι πολύ σημαντικές έχουμε βεβαίως και τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε και νέες διμερείς εμπορικές συμφωνίες για να υπογραμμίσουμε πιο ρητά τη σημασία της βιοποικιλότητας σε σχέση με πολιτιστικά θέματα, αλληλεία, δασοκομεία και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα για εκείνα των ηθαγενών και των τοπικών κοινοτήτων που τακτικά, τακτικά επηρεάζονται αρνητικά από τις παρεμβάσεις σε αυτά τα πεδία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να υποστηρίξει, να υπογραμμίσει διεθνώς τις αρνητικές επιπτώσεις της μη τήρηση, του μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πλαίσια μεταφοράς τεχνολογία, συνεργατικών πλαισίων, ε, οικοεπισήμανσης, οικολογικής επισήμανσης κτλ. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου βιωσιμότητας επίσης δίνουν ευκαιρίες να δούμε τη βιοποικιλότητα στο ανθρώπινο δικαίωμα πέραν των όσων έχουμε συμφωνήσει με χώρες εταίρους. Ώστε να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τονίζει ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όσες περισσότερες ε, ρήτρες ασφαλείας εγγυήσεις γίνεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν και πάρα πολλές ε, μονομερείς επιμέρους πρωτοβουλίες, η κανονισμοί Timber και FLEGT αλλά και πολλά άλλα παραδείγματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το παράδειγμα σε διμερές επίπεδο πλέον με τρίτες χώρες και εδώ είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε τα αρνητικά παραδείγματα, τον αρνητικό αντίκτυπο του μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και, την... και τα διδάγματα και τη γνώση που μπορεί να μεταφερθεί ως προς τις ωφέλειες που μπορούν να απορρέουν από την προστασία της βιοποικιλότητας. Η συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων, η συνεργασία με εξειδικευμένες υπηρεσίες και οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, που συμμετέχουν και διαχειρίζονται καμιά φορά τα μέσα αυτά και της εξωτερικής χρηματοδότησης που ρέει προς τις ε, τρίτες χώρες επί τη βάση των κοινών αρχών και αξιών συμπεριλαμβανομένη της προστασία της βιοπικιλότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μείνω εδώ, αλλά περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ε, ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε περιορισμένη ανεξάρτητη έρευνα προς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις αναγνώρισεις της προστασίας βιοποικιλότητας στο ανθρώπινο δικαίωμα. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, αλλά θα ήταν θετικό πιστεύω να προτείνουμε να ζητήσουμε και άλλες για να ξέρουμε ακριβώς πόσες πρακτικές υποστηρίζουν μία προσέγγιση που να βασίζεται στον άνθρωπο human-based approach, για να το πούμε ελληνικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ιζαμπέλα, στην Άννα. Η Ιζαμπέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ και μας κάνατε την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι έχουμε πλήρη συνέστηση του τι συμβαίνει επί της γης, όλα αυτά, οι φυσικές καταστροφές, όλα αυτά είναι αλληλένδετα, κάτι το οποίο ε, δυστυχώς γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να ε, θίξω ένα σημείο και ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε και παραδείγματα η σχέση μεταξύ κρατών, οι διακρατικές σχέσεις ιδιαίτερα. Μιλήσατε για ανταλλαγές πληροφοριών σε επιστημονικό επίπεδο και ως προς τις κλιματικές αλλαγές και θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα περισσότερα ως προς αυτό το σκέλος. Μιλήσατε για τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις θέλαμε να μας πείτε πού λειτουργεί τι καλύτερα, τι θα πρέπει να προσέξουμε και επίσης εκτιμώ το γεγονός ότι επιμείνατε ως προς την εφαρμογή, γιατί όλα τα κείμενα, όποια και να είναι, αν μείνουν επί χάρτου δεν σημαίνουν τίποτα θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το κανονιστικό πλαίσιο. Ε, εάν θέλετε να μας ε, δώσετε συμβουλές, έχει καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραμείνω μέχρι τέλους. Η Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική αυτή μελέτη και είναι πολύ επικαιρή καθώς όπως είπατε τώρα όλοι μιλάνε για την κλιματική δράση κατά της ε, κλιματικής κρίσης, αλλά η βιοπικιλότητα δεν είναι στο προσκήνιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Η πρώτη είναι η εξή. Η Κομισιόν τον Δεκέμβριο που μας πέρασε ε, εξέδωσε το λεγόμενο πράσινο deal, αλλά δεν το αναφέρετε στην μελέτη σας. Το ερώτημά μου είναι το εξής αν μπορείτε να επεκταθείτε πώς βλέπετε την βιοπικιλότητα ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν θα θέλατε να δείτε κάποια περαιτέρω πρόοδο καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το τελικό έγγραφο. Μετά τονίσατε την έλλειψη αξιόπιστων συστημάτων παρακολούθησης της σχετικής σύμβασης του ΟΗΕ. Έχουμε όμως κάποιους μηχανισμούς για παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίπεδο του ΙΕ. Οπότε το ερώτημα μου είναι κατά πόσο θα μπορούσαμε να ενσωματώνουμε στα διάφορα μέσα την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας. Μετά, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για το κατά πόσο μπορεί να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια για αυτά τα ζητήματα, γιατί είδαμε κάτι σχετικό για το κλίμα. Και μετά αναφέρατε το πρόβλημα με την εξωτερική χρηματοδότηση στην τελευταία διαφάνεια όπου λέτε ότι η εξωτερική χρηματοδότηση καταστρέφει τη βιοποικιλότητα. Έχετε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις με κοινοτική χρηματοδότηση όπου θα μπορούσαμε να δούμε ή να μας εξηγήσετε πώς ε, λειτουργεί κάτι τέτοιο και τι μπορεί να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, αυτό βεβαίω απευθύνεται πιο πολύ σε εμά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθέσει μία μελέτη και μία σχετική έκθεση πρωτοβουλία, ε, το Renew συγκεκριμένα, αλλά δεν βλέπω κάποιον από το Renew εδώ. Και οφείλω να πω ότι δεν μου αρέσει αυτό. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο Νάτσο θέλει το λόγο, όχι. Κάποιος άλλος. Deux questions également. Και εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Μιλήσατε για τις χημικές ουσίες και την στρατηγική σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοπικιλότητα. Ξέρετε ότι υπάρχει νομοθεσία REACH, η οποία είναι ελληματική. Βλέπουμε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας ισχύει μόνο κατά 30%. Δεν ξέρω κατά πόσο δικά σας μέσα μπορούν να κάνουν αυτό τον συσχετισμό μεταξύ της μη εφαρμογής και της στήρησης της βιοπικιλότητας, γνωρίζοντας ότι οι χημικές ουσίες είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως, οι χημικές ουσίες μεταφέρονται, μεταφέρονται και καταναλώνονται και μπορούν να έχουν επιπτώσεις και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχουν γίνει μελέτες επί του θέματος. Επίσης είδαμε σημαντικές εκστρατείες για την εξαφάνιση ζωικών ειδών και ιδιαίτερα ως προς τα θηλαστικά. Ε, έγινε λόγος για τις μέλισσες και μια μεγάλη εκστρατεία, αλλά βλέπουμε ότι αυτό ισχύει και για τα έντομα γενικότερα, δηλαδή πλήττονται και είναι ήδη προς εξαφάνιση. Έχετε συγκεκριμένες υποδείξεις για το κατά πόσο αυτό έχει επιπτώσει στους ανθρώπους, γιατί πολλοί λένε ότι η εξαφάνιση των εντόμων δεν θα έχει επιπτώσεις επί ουδενός. Αλλά αν δούμε τις επιπτώσεις στη γεωργία, στη περιοχή του Σαχέλ βλέπουμε ότι η εξαφάνιση των εντόμων θα είχε μεγάλες επιπτώσεις ε, στη γεωργική παραγωγή. Έχουν γίνει μελέτες επί του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλες αυτές οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για την πρώτη ερώτηση της διακρατικές σχέσεις και πρακτικά παραδείγματα όπου μπορούμε να δούμε ε, τη βιοποικιλότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, νομίζω το καλύτερο παράδειγμα είναι η συνεργασία για την κλιματική αλλαγή. Εδώ πέρα βλέπουμε την περισσότερη χρηματοδότηση, επιστημονική συνεργασία. Ήδη στον τομέα των δασών βλέπουμε πως μπορεί να είναι ένας τομέας όπου ε, υπάρχει σαφώς μία διευθύνση κατεύθυνση που υπάρχει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση περί βιοποικιλότητας, οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε μία προσέγγιση Red Sin. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ε, σχετική κατεύθυνση και νομίζω ότι έχει προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο και στα θέματα κλιματικής αλλαγής, αλλά έχει υπάρξει μικρή αντίδραση συνολικά και ανταπόκριση. Οπότε δουλεύουμε διμερώς με κάποιες χώρες εταίρους ε, που βλέπουν την ε, σημασία αυτή για να μπορέσουν ακριβώς να κάνουν τη διαφορά και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω τώρα που έχουν πλέον αναδειχθεί οι ωκεανοί έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιες ε, θα είναι οι δυνατότητες προσαρμογής ε, των ωκεανών στην κλιματική αλλαγή με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και κοιτώντας βεβαίως την προσέγγιση οικοσυστημάτων που μας ε, προσφέρεται. Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να εξοδευτεί και η σχετική χρηματοδότηση, αλλά και πώς η επιστημονική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τώρα, για το τι γίνεται διμερός. Ε, υπάρχει το σκεπτικό της διαδικασίας όπου ξεκινάμε με την ομοθεσία μιας τρίτη χώρα αντί να επιβάλλουμε τις προδιαγραφές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίω έχουμε τι εθνικέ αντί για τι ε, διεθνεί προδιαγραφέ. Μια συμμετοχική διαδικασία με τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, κοινή παρακολούθηση καθώς και μία ρητή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης η οποία θα μπορέσει να δείξει πώς ακριβώς οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε πολυμερείς ε, διαδικασίες. Όλα αυτά ε, έχουν αναγραφεί σχετική βιβλιογραφία ως πολύ θετικά και υπάρχουν διαφορές προκλήσεις, υπάρχουν πράγματα όμως τα οποία μπορούμε να διδαχτούμε από πρωτοβουλίες σε άλλους κλάδους, τους ωκεανούς, τις ανανεώσιμες για τα θέματα του πράσινου ντύλου. για τον οποίο ε, δεν ε, τον ανέφερε το εξή. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια προσέγγιση η οποία βλέπει τα περιβαλλοντικά ζητήματα μεμονωμένα, δηλαδή έχουμε την κλιματική αλλαγή ασύνδετη με την βιοπικιλότητα και αυτά τα δύο ασύνδετα με τα χημικά, κάτι το οποίο ακριβώς δεν υποστηρίζει το σκεπτικό της ε, πολιτικής συνοχής σε όλα αυτά τα ζητήματα περιβαλλοντικής συνεργασίας. Επίσης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, υπήρχε ελάχιστη έπαφη με ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων είτε της βιοπικιλότητας και νομίζω ότι τώρα υπάρχει ευκαιρία που οριστικοποιείται η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκαθαρίσουμε νομίζω την σημασία της βιοπικιλότητας για άλλους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και η δυνατότητα να δούμε αυτούς τους τομείς μέσω κάποιων προσεγγίσεων ε, τις οποίες ήδη έχουμε συμφωνήσει και που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή αυτό σχετίζεται και με αυτό το οποίο είπαμε για τα χημικά. Γνωρίζω πως οι ΜΚΟ ζητάνε περισσότερη προσοχή στην σχέση μεταξύ χημικών και βιοποικιλότητας. Δεν είναι μια σύνδεση η οποία έχει ήδη ε, γίνει. Η νέα στρατηγική για την βιοπικιλότητα υπάρχει και είναι και ένα πολύ τεχνικό ζήτημα, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι οι ευρύτερε συνέπειε, ειδικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά σε άλλες χώρες, ε, δεν είναι στο προσκήνιο, αλλά οπωσδήποτε αυτές είναι οι συνέπειες ε, που έχουν οι περιορισμένες ε, πρόοδοι που υπάρχουν στον τομέα αυτής της νομοθεσίας. Οπωσδήποτε αυτό το οποίο τεθεί για το πώς τα στοιχεία παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να επηρεάσουν είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ανέφερα ήδη την έκθεση για να τονίσω ότι μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά εάν η συνολική αυτή αναθεώρηση και τα άλλα υφιστάμενα μέσα για την αξιολόγηση ε, θα μπορούσαν να ενσωματώσουν κάποιες ανησυχίες για την βιοπικιλότητα. Οπωσδήποτε βλέπουμε κάποια αλλαγή από όταν έχει γίνει πολύ βασική κλιματική αλλαγή στα θεσμικά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και πάλι δεν πρέπει να το δούμε απομονωμένο το ζήτημα αυτό από τα άλλα. Και ίσως κάποιοι συνάδελφοι θα μπορούσαν ακριβώς να δουν την υφιστάμενη κατεύθυνση που υπάρχει σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να την εφαρμόσουν και στο ζήτημα της ε, βιοπικιλότητας. Ακριβώ ε, για να ενωθούν αυτές οι δύο κοινότητες ε, βιοπικιλότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις αναψώμενες χώρες. Τώρα δεν έχω συγκεκριμένα παραδείγματα για την αρνητική επίπτωση της ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση υδροηλεκτρικών έργων ή έργων Red Sin ή έργων δασοκομείας που είχαν πολύ σοβαρές ε, αμφιβολίες για την επίπτωσή τους ε, στους αυτόχθονες πληθυσμούς και ακριβώ ε, έχει υπάρξει ένας κατάλογος ε, αυτοχθόνων ε, πληθυσμών που σχετίζονται με την προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Οπότε πρέπει να διασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση για να διασφαλίσουμε και τα σχετικά ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Τέλος, για την απώλεια των ειδών. Εδώ πέρα έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα ζητήματος το οποίο θεωρούσαμε περιθωριακό, προστασία των πάντα ή πράγματα που είναι προβλήματα πολυτελείας. Ε, βλέπουμε όμως πως ε, η απώλεια των επικονιαστών και των μελισσών επηρεάζει την ε, διατροφική ασφάλεια ή τα ζώα που χάνονται και είναι στην κορυφή της ε, τροφικής αλυσίδας ε, ε, κατά κάποιον τρόπο παρέχουν υπηρεσίες και η απολυά τους μπορεί να έχει πολύ σοβαρέ συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή ή στα τρόφιμα και στο νερό. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς μιλήσατε για ένα συγκεκριμένο είδος Μιλήσατε για διμερείς σχέσεις με χώρες γνωρίζοντας ότι η νομοθεσία ξεκινάει από το σημείο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν παράνομοι ε, θύλακες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ε, προωθήθηκε αυτή η νομοθεσία με εμπορικές σχέσεις σε σχέση με τα δάση. Δηλαδή δεν πρόκειται ε, για ε, νομοθεσία απαγόρευσης, απλώς επιτρέπει στις χώρες αυτές να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη νομοθεσία. Μιλάμε για ένα πλαίσιο, ε, εθελοντικό πλαίσιο, μια εθελούσια βάση και ε, εκούσια διαβήματα. Θεωρείτε ότι η ΦΛΕΚΤ ε, είναι κάτι το θετικό γιατί διαφορετικά φτάνουμε στην πλήρη απαγόρευση. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο αυτό το εκούσιο πλαίσιο λειτουργεί, γιατί οι μελέτες μας δείχνουν ότι δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχουν γίνει έρευνες. Άννα, θέλεις και εσύ να ρωτήσεις κάτι. Ναι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο, ε, στην Επιτροπή είχαμε σκεφτεί να συντάξουμε μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία σχετικά με τη σχέση βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, εσωτερικό έγγραφο ενδεχομένως, αλλά θέλαμε να ε, ε, συσχετίσουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική αλλαγή. Ποιε βασικές πτυχές υπάρχουν ή θα μας προτείνατε και θεωρείτε ότι είναι μια ορθή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, το ΦΛΕΚ ξεκίνησε ως εθελοντική πρωτοβουλία, μετά ήρθε και το νομικό πλαίσιο για τα δάση. Υπάρχει ένα φάσμα ή ένα συσχετισμός ε, προσφοράς κινήτρων μονομερών και πολυμερών πρωτοβουλειών νομίζω ότι μέσω του FLEGD η πρόσβαση στην αγορά δημιούργησε μια πολιτική βούληση αλλά χρειάζεται και μια γνήσια βούληση κοινών προσεγγίσεων και κοινή μάθησης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε και παραδείγματα στη βιβλιογραφία και από την κοινωνία των πολιτών και από χώρες εταίρους που έχουν χαιρετήσει την προσέγγιση αυτή και που δημιούργησαν μια πίεση για να υπάρξει δράση. Αυτός είναι ο πολιτικός κίνδυνος, αλλά εφόσον οι προϋποθέσεις της πρόσβασης στην αγορά βασίζονται σε πολυμερείς στόχους και μια προσέγγιση που αφορά και στους εταίρους, αυτό έχουμε μάθει, φαίνεται ότι λειτουργεί. Τώρα, πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερη προσοχή διεθνώς στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία της φύσης ή στο κλίμα. Υπάρχουν ευκαιρίες, ευκαιρίες εντός της κλιματικής αλλαγής να δει κανεί τη βιοποικιλότητα στο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτά τα έχουμε συμπεριλάβει και στην έκθεση σε σχέση με τα δάση, τους ωκεανούς, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κρίσεων. αλλά υπάρχει και το πεδίο της ε, σχέσης μεταξύ βιοποικιλότητας και χημικών, χρήσης χημικών, τη σχέση με την ανθρώπινη, με τη δημόσια υγεία, την ε, μεγάλη σημασία της βιοποικιλότητας για τα δικαιώματα των παιδιών, στοιχεία που δεν θα ενέπιπταν δηλαδή αναγκαστικά και πιστεύω ότι είναι ένα κέριο χρονικό σημείο για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτά θα μας επιτρέψουν πράγματι να λάβουμε υπόψη σας ε, τα σχόλιά σας στη δουλειά που έχουμε να κάνουμε εφόσον υπάρξει συμφωνία γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση για την Υποεπιτροπή Δικαιωμάτων λοιπόν και τη σχέση με την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας και θα περάσουμε στο σημείο 5 λέει η Πρόεδρος δεν ξέρω αν ο κύριος Γεουντά Σαουντ είναι παρόν, τότε απλώς να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 4 παρακαλώ. On va commencer notre point 5, euh, qui est un échange de vues. Φτάνουμε στο σημείο 5 που προβλέπει μια ανταλλαγή απόψεων με το Γεχούντα Σόλ, συνειδητή της, ε, σπάζοντας, της οργάνωσης σπάζοντας τη σιωπή είναι ο ιδρυτής της οργάνωσης Σπάζοντας τη Σιωπή. Είσαστε συνομιλητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και χρόνια. Όταν επισκεφθήκατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και όταν επισκεφθήκαμε εμείς το Ισραήλ. Ήσασταν στον τελικό κατάλογο για το βραβείο Ζαχάροφ εδώ και λίγα χρόνια. Νομίζω ότι γνωρίζετε την οργάνωση σπάζοντας τη σιωπή που απαρτίζεται από πρώην στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού που υπηρέτησαν στα κατεχόμενα. Θα μας μιλήσετε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το κομμάτι του κόσμου, ε, πρόκειται για πολύ δύσκολη κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να ακούσουμε όλους τους συνομιλητές που γνώρισαν δύσκολες καταστάσεις ως προς την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να πω ότι μία παρόμοια οργάνωση είναι ευεργετική για τα δημοκρατικά δικαιώματα και για την πρόθεση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρω ότι πολύ συχνά ήταν πολύ δύσκολο για την οργάνωσή σας να δράσει ιδιαίτερα στο Ισραήλ αλλά και στα κατεχόμενα. Περιμένουμε λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε γιατί στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκείνους οι οποίοι ε, στην ουσία ε, προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά περίπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας σήμερα και για την ευκαιρία να έχουμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Για Χούντα Σαούλ λέγομαι. 37 ετών γέννημα θρέμα της Ιερουσαλήμ και της δεξιάς στο Ισραήλ. Πήγα σχολείο σε έναν οικισμό στην Δυτική Οχθή. Τα αδέρφια μου οικίζουν σήμερα, οπότε ιδεολογικά από εκεί καταγούμε. Τελείωσα το σχολείο, πήγα στρατό τρία χρόνια. Παίζει κατατάχθηκα γιατί σκέφτηκα ότι είχε φτάσει η στιγμή της δικής μου γενιάς για να υπερευστεί την πατρίδα μας ε, επί Ιντιφάντας τότε. Όταν τελείωσα όμως την εκπαίδευσή μου και έφτασα στα κατεχόμενα, πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι πολλά, τα περισσότερα πως έκανα, είχαν στόχο να διατηρήσουν την ε, απόλυτη στρατιωτική κυριαρχία μας επί ολόκληρου του Παλαιστινιακού πληθυσμού και άρχισαν να ανακύπτουν διάφορα ερωτήματα. Το... Η ένταξή μου στην οργάνωση αυτή ήταν αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία. Ένα από αυτά τα οποία κάναμε ω στρατιώτε στα κατεχόμενα είναι αυτό το οποίο λέμε ε, να κάνουμε αισθητή την παρουσία μα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτή τη φράση. Ε, το σκεπτικό είναι το εξή αν οι Παλαιστίνοι έχουν την αίσθηση ότι ο στρατός είναι ανα πάση στιγμή παντού, θα φοβούνται να επιτεθούν. Οπότε τι κάνουμε γι' αυτό, κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Σε διάφορα μέρη της Δυτικής Όχθης ε, εμφανιζόμαστε με διάφορους τρόπους. Στην ε, Χεβρώνα που υπηρέτησα πάνω από ένα έτος, τη μεγαλύτερη ε, Παλαιστινιακή πόλη στην Δυτική Όχθη πέρα από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κάναμε το εξή. Είχαμε περιπολίες ε, το 24ωρο, η νυχτερινή βαριά ήταν 10 με 6, 8 ώρο, περπατάμε στους δρόμους της ε, παλιάς ε, πόλης, μπαίνει σε ένα σπίτι, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες. Ένα σπίτι τυχαίο. Ένας λοχείας επικεφαλής επιλέγει τα σπίτια, ξυπνά στην οικογένεια, ψάχνεις το σπίτι, φαντάζεστε τι συμβαίνει όταν μπει ο στρατός στο σπίτι σου 3 ώρα το πρωί. Ε, Βεβαίω, αυτό που έχουμε συνηθίσει εμεί ε, στις δημοκρατικές χώρες, για να μπει κάποιο ε, στο σπίτι σου, πρέπει να υπάρχει μια υποψία, ένα ένταλμα που έχει υπογράψει δικαστής και τα λοιπά. Αυτά δεν υπάρχουν στα κατεχόμενα. Όλα αυτά είναι νόμιμα σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο. Επιλέγουμε τυχαία ένα σπίτι, μπαίνουμε μέσα, ξυπνάμε την οικογένεια, ψάχνουμε Βγαίνουμε στον δρόμο, βαράμε πόρτες, κάνουμε θόρυβο. Αυτός είναι, αυτή είναι η φύση της ε, στρατιωτικής κατοχής. Σαν δικτωρία κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τελειώνει η έρευνα του σπιτιού, βγαίνουμε στον δρόμο, πηγαίνουμε στη γωνία ενός άλλου δρόμου, μπαίνουμε σε ένα άλλο σπίτι, ξυπνάμε άλλη μια οικογένεια, ψάχνουμε το σπίτι, ξαναβγαίνουμε, ανεβαίνουμε στην ταράτσα, από τη μία ταράτσα στην άλλη, την επόμενη. Ε, είναι 8 ώρες βάρδια έτσι από τον Σεπτέμβριο του 2000 ε, ε, για ένα χρόνο δεν σταμάτησε καθόλου. Το σκεπτικό είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να νιώσουν οι Παλαιστίνοι ότι ο στρατός είναι παντού. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αυτό το οποίο λέμε στον στρατό ε, να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι τους κυνηγάνε εντός ε, του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Γιατί βεβαίω ο μόνος τρόπος να τους ε, διοικούμε παρά τη θέλησή τους στα κατεχόμενα είναι ο και όταν ε, συνηθίσουν ένα επίπεδο φόβου το αυξάνεις και τα λοιπά χωρίς τέλος. Και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να εκφοβήσουμε τον Παλαιστινιακό πληθυσμό, να τσακίσουμε την Παλαιστινιακή κοινωνία για να μην μπορούν να μας προκαλέσουν. Φτιάχνουμε οικισμούς για να μην αναπτυχθεί ποτέ Παλαιστινιακή κυριαρχία. Αλλά η κατοχή δεν παραμένει στα κατεχόμενα μόνο. Ε, η κατοχή επεκτείνεται και στο Ισραήλ σιγά σιγά. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε υπουργούς, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να επιτίθενται ουσιαστικά σε οποιονδήποτε αμφισβητεί την πολιτική στα κατεχόμενα. Οι υπουργοί που λένε τη δικιά μας οργάνωση, οι προδότες, κατάσκοπους κτλ. Η Μπιτσέλε, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού μίλησε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, η κυβέρνηση είπε να τους αφαιρεθεί η υπηκότητα. Και δεν είναι μόνο η κοινωνία των πολιτών. Ο Υφυπουργό Άμυνα μία μέρα πρότεινε να βάλει μία μπουλντόζα και να κατεδαφίσει το ανώτατο δικαστήριο. Γιατί το ανώτατο δικαστήριο έβγαλε μία απόφαση για έναν οικισμό που δεν του άρεσε. Αλλά δεν είναι μόνο. Δεν μένουν μόνο στα λόγια μια γκαλερί στην Ιερουσαλήμ κλείνει αυτές τις μέρες ε, από τον ε, Δήμαρχο της Ιερουσαλήμ επειδή μας φιλοξένησε για μια εκδήλωση. Ο πρώην υπουργό ε, Παιδείας πέρασε από το Βουλή ένα νόμο που λεγόταν ο νόμος σπάζοντας την σιωπή και δίνει στον Υπουργό την δυνατότητα να δημιουργήσει μια μαύρη λίστα οργανώσεων που απαγορεύεται να πάνε στα σχολεία. Οπότε τώρα θα παρακολουθείτε το τι λέει ο καθένα ανάλογα με το, τις απόψεις του Υπουργού. Λοιπόν, η ιδέα που είχαμε επί δεκαετίες ότι το Ισραήλ θα μπορεί να διατηρεί μια κατάσταση ενός κράτους με δύο καθεστώτα, δηλαδή μια δημοκρατία εντός ε, της πράσινης γραμμής και στη στρατιωτική δικτατορία στα κατεχόμενα, χωρίς το ένα να επηρεάζει το άλλο, ε, αυτή η ιδέα καταραίει. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Ισραηλινή πολιτική προχωρά. Δεν είναι το θέμα μόνο πλέον η κατοχή, μιλάμε για προσάρτηση. Δεν μιλάμε ότι γίνονται μόνο τα προσωρινά μόνιμα, ούτε μιλάμε για προσάρτηση εδαφών. Μιλάμε απλά για εδάφη τα οποία καταλαμβάνουμε δια της βίας ε, και ενάντια στο διεθνές παίρνουμε την επικράτεια και αφήνουμε τους Παλαιστινίους χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Και ουσιαστικά δημιουργούμε ένα ε, Ισραηλινό apartheid, κάτι στο οποίο θα έπρεπε να είμαστε όλοι εναντί. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ που έρχεται. Το σχέδιο του Τραμπ, κατά την άποψή μου, είναι μια προσπάθεια να δοθεί διεθνής νομιμοποίηση σε αυτά τα οποία περιέγραψα. Να εδρεωθεί δηλαδή ο μόνιμος Ισραηλινός έλεγχος επί των Παλαιστινίων χωρίς να έχουν οι Παλαιστινοί κυριαρχία και αυτοδιάθεση. Να παίρνουμε κομμάτια γης ε, κατακαιρματισμένα με γύρω-γύρω ε, Ισραηλινή ε, γη με Ισραηλινούς δρόμους με την Ανατολική Ιερουσαλήμ να πηγαίνει στο Ισραήλ, ουσιαστικά παραβιάζοντας την διεθνή συνένεση και προσπαθώντας να εδραιώσουμε ε, μόνιμο έλεγχο του Ισραήλ ε, επί των Παλαιστινίων. Και αυτό το λέμε ειρήνη, που είναι το χειρότερο. Λοιπόν, ε, μην έχετε καμία αμφιβολία. Είμαι σιωνιστής. Θεωρώ ότι ε, πρέπει να έχουν αυτοδιάθεση οι Εβραίοι από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη θάλασσα και μπορώ να, θα πεθάνω γι' αυτό. Αλλά δεν δέχομαι ότι ο μόνος τρόπος που εμείς ε, οι Εβραίοι θα έχουμε αυτοδιάθεση είναι να μην έχουν αυτό το δικαίωμα οι Παλαιστίνοι. Η άποψη αυτή και η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο ανήθικη, αλλά απειλεί την νομιμοποίηση του κράτους του Ισραήλ. Ο Τραμπ ή μάλλον θα έλεγα γι' αυτό θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ. Η μόνη διέξοδος είναι ε, να φύγουν και οι δύο πλευρές από το δωμάτιο με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει το σχέδιο Τραμπ. Όταν περπατούσα στους δρόμους της Δυτικής Όχθης ως στρατιώτης και έμπαινα σε σπίτια με στη μέση της νύχτας για να τους δημιουργήσω την αίσθηση ότι είναι κυνηγημένοι. Πολιτικά αυτό το οποίο έκανα και αυτό το οποίο κάνει η κατοχή μας ε, είναι να έχει ως στόχο την παράδοση των Παλαιστινίων. Αυτός είναι και ο πολιτικός στόχος του σχεδίου Τραμπ. Δεν επιτυγχάνει την ειρήνη, αλλά προσπαθεί να επιτύχει την παράδοση των Παλαιστινίων. Γι' αυτό το απορρίπτουν οι Παλαιστινοί. Και δικαίως δεν είναι συνταγή για ειρηνή, είναι συνταγή για μόνιμες συγκρούσεις και βία. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το απορρίψετε αυτό το σχέδιο. Εμείς, Ισραηλοί και Παλαιστίνοι, αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον, όχι το μέλλον που σχεδιάζει για εμάς ο Τραμπ. Και ελπίζω να κάνετε ό,τι μπορείτε, έτσι ώστε η γραμμή Τραμπ να μην αποτελέσει τη νέα βάση διαπραγματεύσεων, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μόνιμη σύγκρουση, αλλά να απορριφθεί εντελώ. Και να έχουν αξιοπρέπεια και δικαιώματα και οι Ισραηλοί και οι Παλαιστινοί. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε Γεχούντα. Τώρα, ποιος θα ήθελε να μιλήσει, ο κύριος Βαντάλεν και Νάτσο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κοιτάω τι συμβαίνει αυτή την στιγμή. Ενώ δεν ξέρω ποιος προσκάλεσε τον κύριο. Εγώ δεν έλαβα την πρόσκληση ούτε την απάντησα αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα είναι μία από τις ελλείψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία από τις ελλείψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η έλλειψη αντιλόγου, λόγου και αντιλόγου. Και μία από τις ελλείψεις αυτού του Κοινοβουλίου είναι το ότι συνεχώς ακούγονται διάφορες θέσεις χωρίς να υπάρχει χώρος για απόχρωση και διάλογο. Έρχεται εδώ πέρα ο κύριος αυτός, βγάζει ένα λόγο επί τρία λεπτά, απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ, όπως το λέει, αλλά που είναι ο αντίλογος. Ακούσαμε τη μία πλευρά. Δεν ακούστηκε τίποτα διαφορετικό και δεν ακούστηκε καμία απόχρωση. Γιατί αγαπητέ κύριε Σαουλ, θα ακούγαμε σε αυτή την περίπτωση και τα εγκλήματα της Χαμάς στα κατεχόμενα που έχει στην λωρίδα της Γάζας τους κυβερνάει εκεί πέρα με το κνούτο και δεν ακούω να λέτε τίποτα οπότε πρόκειται για μια λυπηρή στιγμή έχουμε μια τελείως μονόπλευρη παρουσίαση και εγώ θεωρώ ότι είναι εκπληκτικό όμω ότι έχει τόσο φοβερή δημοκρατία το Ισραήλ ώστε επιτρέπεται να λέτε αυτά τα πράγματα. Αν τα κάνατε αυτά στη Σαουδική Αραβία ή την Ιεμένη, το Πακιστάν, τη Βενεζουέλα ή το Ιράν, το Κονγκό, το Αφγανιστάν. Ε, λέω συγκεκριμένα τις χώρες αυτές γιατί είναι χώρες που είναι στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έτσι. λοιπόν δεν θα είχατε αυτήν την ε, δυνατότητα. Αλλά δεν είναι σωστό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούγεται λόγος ε, χωρίς ε, αντίλογο. Και εγώ θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρωτού κάνω την ερώτησή μου, ήθελα να σχολιάσω ε, τα όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Δεν είμαστε στην Επιτροπή Εκτορικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είμαστε. Καλούμε ανθρώπους που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε και ορισμό για τον υπερασπιστή των δικαιωμάτων. Κάποιο που δεν χρησιμοποιεί βία, που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρί να παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Νομίζω ότι μπορούμε να προσκαλούμε και στο μέλλον Άλλου ανθρώπου τη ίδια περιοχή που μπορεί να έχουν μια άλλη προσέγγιση, αλλά ω μέλο τη επιτροπή πολύ χαίρομαι που ήρθατε εδώ και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για, τα, για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε και για τα ευγενικά σα λόγια. Ένα από του λόγου που είμαι ικανοποιημένη για την παρουσία σα είναι και ο εξή και κάνω την ερώτησή μου. Οι φωνέ υπέρ της ειρήνης και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη έχουν σιγάσει αυτή τη στιγμή. είναι όλο και λιγότερες. Σε όποια πλευρά και να με όποια πλευρά και να συντάσσεται κανείς, χρειάζεται μία λύση ειρήνευσης και επομένως είναι πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθεί να υποστηρίζει και να υποστηρίζει περισσότερο θα έλεγα όλους εκείνους τους φορείς και τις οργανώσεις που δουλεύουν υπέρ της ειρήνης στην περιοχή. Επομένως κύριε Σαούλ, και εδώ τοποθετούμε λίγο περισσότερο σε διεθνέ επίπεδο. Μιλάτε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι και αυτοί που μαρτυρούν οτιδήποτε που καταδίδουν, που καταγγέλνουν αυτά τα φαινόματα αντιμετωπίζονται δεινά. Η δική σας οργάνωση έχει σχέσεις με άλλες οργανώσεις, άλλους φορείς που ασχολούνται με το ίδιο θέμα και που καταγγέλουν. Και τώρα για να επανέλθω στο διεθνές πλαίσιο, επικρίνεται το σχέδιο, πλάν, το σχέδιο Τραμπ, με συγχωρείτε, και αντιλαμβάνουμε την κριτική σας. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό και ένα από τα επιχειρήματα που ακούστηκα ήταν ότι ναι, ναι, επικρίνουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και καλύτερο σχέδιο να προτείνει. Τι κατά την γνώμη σας θα ήταν ένα καλύτερο σχέδιο ώστε να επιληθεί ένα πρόβλημα που θέλουμε όλοι να επιληθεί. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ινσύρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να καλωσορίσω τον ομιλητή μας ε, Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Σας είχα δει νομίζω τον Αύγουστο όπου κάποια μέλη διαφόρων πολιτικών ομάδων επισκεφθήκαμε το Ισραήλ και την ε, Παλαιστίνη. Και είχαμε συναντηθεί στην Ιερουσαλήμ μεταξύ άλλων. Καθυστέρησα και ίσως ήδη να αναφερθήκατε σε αυτό που θέλω να ρωτήσω, αλλά ήθελα να υπογραμμίσω και το θέμα του σχεδίου Τραμπ. Πολλοί εξημών που πιστεύουν σε μια λύση δύο κρατών με δύο δημοκρατικά κράτη που θα συνεπάρχουν ειρηνικά, για αυτούς τους ανθρώπους η πρόταση Τραμπ, το αφήγημα Τραμπ ήταν ε, καταθλιπτικό. Γιατί λαμβάνει υπόψη του μόνο τη μία πλευρά και καθόλου την άλλη. Τώρα σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Ποια είναι η αποψή σας για τις εκλογές αυτές, για την αντιπαράθεση αυτή, μήπως υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Μήπως υπάρχει κάποια ελπίδα για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, για μια περισσότερη πιθανότητα για λύση δύο κρατών. Ευχαριστώ, Νάτσο. Ευχαριστώ Μαρία, θα μιλήσω ισπανικά. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω για την τοποθέτησή σας και τη δουλειά σας για τα όσα είπε ο κύριος Βαντάλεν, ο συνάδελφος. Εκφράζει την απόψή του βεβαίως. Και όλοι έχουμε επαρκή εμπειρία και γνώση για να γνωρίζουμε ότι η δική σας άποψη δεν είναι το σύνολο των απόψεων ή το θέμα. Εγώ όμως σας ευχαριστώ που εκφράζετε την άποψή σας και για τη δουλειά που κάνει η οργάνωσή σας. Αναφερθήκατε σε μια εποχή, σε μια περίοδο που είχαμε πολύ μεγάλη ένταση και βία. Αλλά τελικά αυτό που με ανισχύει εμένα είναι ότι επικρατούν τα αφηγήματα των άκρων από κάθε πλευρά. κανείς έχει την τάση να υποστηρίξει τη γραμμή του Ισραήλ γιατί είναι μια δημοκρατία, μια δημοκρατική χώρα και έχουμε όλοι βέβαια προβλήματα με την εύρυθμη δημοκρατία και στις χώρες μας αλλά δεν υπάρχουν αποχρώσεις ε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να υπερασπιστεί κανείς καμία τοποθέτηση άποψη που να προέρχεται από την Παλαιστίνη και φαίνεται σαν να λείπουν γέφυρες, σαν να λείπουν κοινοί τόποι, κοινά σημεία. Ενώ αντίθετα θα πρέπει σε αυτό το κοινό έδαφος να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε. Γιατί αν συνδυάσουμε τις ακρότητες της τοποθέτησης της μίας και της άλλης πλευράς δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, καμία ελπίδα. Πρέπει πάντως πάση θυσία να διατηρήσουμε εν ζωή την ελπίδα, την ιδέα των δύο κρατών. Και οποιαδήποτε απόπειρα, οποιασδήποτε άλλης δύναμης δεν συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή και το σχέδιο του Τραμπ σίγουρα δεν συνεισφέρει, δεν θα συνεισφέρει και δεν θα βοηθήσει. Και έχοντας πει αυτά, εσείς πιστεύετε ότι μια επιφανέστερη διεθνής αναγνώριση. Επίσημη αναγνώριση της Παλαιστινιακής Αρχής ως κρατική οντότητα από περισσότερες χώρες στον κόσμο θα βοηθούσε. Γιατί δεν αναφερθήκατε συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα, ε, θα με ενδιαφέρει πολύ να τα ακούσω. Σας ευχαριστώ. Σαλίμα. ευχαριστώ. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος της ομάδας μου. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι υπερήφανη διότι σας είχαμε προτείνει για το βραβείο Ζαχάροφ. Τώρα, ε, δεν θα ήθελα να προσθέσω πολλά στις ε, ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί. Δύο ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για την καθημερινότητά σας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά. Τι υποστήριξη έχετε από τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και πώς ε, βλέπετε την υποστήριξη από το εξωτερικό για αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο. Επίσης είπατε για πολλές ε, ΜΚΟ που ε, αποτελούν εφεδρικές δυνάμεις στο στρατό του Ισραήλ και μιλάτε για επιθέσεις που έχετε δεχτεί από αυτές τις ΜΚΟ. Πώς τις αντιμετωπίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τις επιθέσεις επιθέσεις που έχετε υποστεί. Και εγώ θα ήθελα να σας υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Καταρχήν είδαμε και μιλήσαμε για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την θέση των ΜΚΟ από το Ισραήλ που μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα και στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα. για ότι ε, δεν μιλήσαμε τόσο πολύ για τους ε, Άραβες που ζουν στο Ισραήλ και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι ΜΚΟ του Ισραήλ επικρίνουν την ε, κυβέρνηση και έχουν ένα ολοένα συρρυκνούμενο χώρο έκφραση. Μιλήσατε για την Μπετσελέμ για την ε, σπάζοντας τη σιωπή και για άλλες οργανώσεις, άλλες μικιό. Θεωρείτε ότι πραγματικά συρρυκνώνεται αυτός ο χώρος ελεύθερης έκφρασης στο Ισραήλ. Δεύτερον, έχουμε λάβει πληροφορίες από παλαιστινιακές πηγές και βλέπουμε ότι υπάρχουν μικιό από πλευράς ε, Παλαιστίνης που δυστυχώς έχουν όλο ένα και μικρότερο χώρο έκφρασης, κάτι το οποίο φυσικά επικρίνουν οι Παλαιστίνοι και η Παλαιστινιακή Αρχή επίσης δεν μπορεί να εκφραστεί τόσο όσο στο παρελθόν. Το νιώθετε και εσείς αυτό και υπάρχει κάποια πλατφόρμα των ΜΚΟ Ισραηλινών και Παλαιστινίων που δίνουν κοινή μάχη για ελεύθερη έκφραση γιατί σήμερα είστε εδώ παρόν γιατί σήμερα ως Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σας δίνουμε το δικαίωμα λόγου. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Βαντάλεν όταν αναφέρει ότι πρέπει να δίνουμε πάντα το λόγο στους άλλους. Είχαμε καλέσει και άλλες μικιό επικριτικές προς την εξουσία, όποια μορφή εξουσίας, άρα δεν μπορεί το ΕΛΚ να μας κατηγορεί ότι δεν δίνουμε το λόγο στους άλλους. Μας διακατέχει η ίδια λογική. Δίνουμε το λόγο στους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από όπου και να προέρχονται, είτε είναι Παλαιστίνοι είτε Ισραηλινοί. Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τους Παλαιστίνιους, ο χώρος τον οποίο, τον οποίο μέρα με τη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσω να καλύψω το εύρος των ερωτήσεων. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον. Υπάρχει αυτή η τάση της συρρήκνωσης του χώρου ελεύθερης ε, έκφρασης υπάρχει βεβαίως ισχύει ως προς την ε, Μπετσελέμ και την ε, σπάζοντας τη σιωπή. Εδώ το βλέπουμε τα τελευταία πέντε χρόνια όπου οι κυβερνήσεις γίνονται όλο και πιο δεξιές και φτάνουν και στην ακραδεξιά. δεξιά. Βλέπουμε ότι υπάρχει επίθεση κατά του οποιοδήποτε επικρίνοντα που επικρίνει επικισμούς. Επίσης υπάρχει ε, και ένα κίνημα κατά τον ΜΚΟ, κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές ε, ΜΚΟ στην ουσία συντονίζουν εκστρατείες για να προωθηθεί νέα νομοθεσία. Αυτό το βλέπουμε. Ως προς τις ε, καθημερινές προκλήσεις, θα σας δώσω ένα παράδειγμα ενός συναδέλφου τις τελευταίες μέρες. Ονομάζεται Ιντο. Είναι επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ισραήλ, με σεμινάρια, συζητήσεις, πάνελ και οδηγεί τους ανθρώπους επιτόπου για να δουν την πραγματικότητα στα κατεχόμενα με χιλιάδες Ισραηλινούς παρόντες και αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Είναι και δάσκαλος και προσπαθούν να τον απολύσουν. Γιατί πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην οργάνωση σπάζοντας τη σιωπή και να είναι και δάσκαλος. Είναι προδότης, δεν μπορεί να είναι δάσκαλος. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μία εκστρατεία κατά του ανθρώπου αυτού, στο σχολείο του στο πρόσωπό του. Πράγματι, οι Παλαιστίνοι εταίροι μας υφίστανται ε, πιέσεις όχι μόνο από το Ισραήλ, αλλά και από την Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και θα ήταν σκόπιμο να έχετε και έναν Παλαιστίνιο εκπρόσωπο να σας μιλήσει για τις προκλήσεις που γνωρίζουν οι Παλαιστίνοι από πλευράς Ισραηλινών αρχών, αλλά και από την Παλαιστινιακή αρχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει να το αμφισβητήσουμε. Είναι ένα θέμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητα παρέμβασης. Συμφωνώ με το εξής. Κάτι το οποίο μας ενοχλεί περισσότερο είναι ε, ότι υπάρχει αυτός ο διεισμός όταν μιλάμε για Ισραήλ και Παλαιστίνη θα πρέπει κανείς να ταχθεί υπέρ των μεν ή των δε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός υπέρ αυτών που είναι ε, ως προς αυτούς που είναι υπέρ της βίας και της τρομοκρατίας και κατά αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μην επιτρέψετε τη συνεχή στρατιωτική δράση του Ισραήλ, να μην γίνει το κράτος του Ισραήλ ένα κράτος apartheid. Ως προς την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, αν γίνει θα βοηθήσει, βεβαίως και θα βοηθήσει. Εάν πιστεύετε στην ύπαρξη δύο κρατών, και Εάν αναγνωρίζουν ε, οι Παλαιστίνοι το Ισραήλ, τότε θα πρέπει να υπάρξει και Ισραηλινό κράτος. Βεβαίως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους Παλαιστίνιους γείτονες. Δεν θα πρέπει να έχει δικαίωμα άρνηση κυρία στο Ισραηλινό κράτος για το αν έχουν δικαίωμα σε κράτος οι Παλαιστίνοι. Αυτό είναι παράδεκτο. Θα αλλάξουν τα πράγματα επιτόπου. Μερικά ναι, μερικά όχι. Ας δούμε το σχέδιο Τραμπ, για παράδειγμα. Αν δούμε την κυβέρνηση Νετανιάχου, βλέπουμε και μερικές άλλες κυβερνήσεις πριν από αυτήν, βλέπουμε ότι το θέμα δεν ήταν οι διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε σε δύο κράτη. Απλώς ε, θέλαμε ε, να φτάσουμε σε ένα αφήγημα όπου θα υπάρχει Ισραηλινικό κράτος και κάτι λιγότερο από Παλαιστινιακό. Θυμάμαι ένα, ένα άρθρο που διάβασα του Νάταν Έσελου, ο οποίος ήταν ε, επικεφαλής σύμβουλος του ε, Νετανιάχου και δημοσίευσε ένα άρθρο αφού συναντήθηκε ο Νετανιάχου με τον Τραμπ στις αρχές Φεβρουαρίου και αναφερόταν το εξής. Ε, σας, σας το αναφέρω από μνήμης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε το θέμα των δύο κρατών στην χτεσινή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι η σωστή λύση. Αυτό λέει ο αρθρογράφος. Το να λέμε ότι οι Παλαιστίνοι ε, αξίζουν να έχουν κράτος πριν από τις διαπραγματεύσεις δεν αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης. Και νομίζω ότι με αυτή τη δήλωση ο Νάταν Έσελ μας, ε, λέει, μας προβάλλει το αφήγημα της Ισραηλινής κυβέρνησης ότι δεν θέλουμε δύο κράτη, θέλουμε να ελέγχουμε τους Παλαιστίνιους με το δικό μας τρόπο και το ζήτημα είναι πόσος θα είναι αυτός ο έλεγχος μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης. Γι' αυτό θεωρώ ότι η αναγνώριση είναι ε, απαράμιλη ανάγκη και βασίζεται και στην πράσινη γραμμή. Και θα σας πω και έναν άλλο λόγο, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Εάν η πραγματικότητα του ενός κράτους που ζούμε εδώ και μισό αιώνα προσπαθήσει να ε, ανυψώσει την πράσινη γραμμή, στην ουσία θέλει να ελέγχει τους Παλαιστίνιους διαπαντός. διαπαντός. Εάν υπάρχει αναγνώριση της πράσινης γραμμής, το θέμα είναι διαφορετικό. Το βασικό που έχετε να κάνετε είναι ε, να πάρετε ε, ένα χαρτί και μολύβι και να ξαναορίσετε την πράσινη γραμμή. Να πρασινίσετε το χάρτη δηλαδή. Ένα κυρίαρχο Παλαιστίνιο κράτος δίπλα στο Ισραήλ όχι το θέμα της Χαμάς. Το αντίθετο. Δύο κράτη, όχι αυτό που θέλει η Χαμάς. Το ίδιο αφορά και την ε, αρχή της διαφοροποίησης. Εσείς οι Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει να συνεισφέρετε στους επικισμούς, στον, ε, στη συνέχιση του ελέγχου των Ισραηλινών στη, στα κατεχόμενα με τους συνεχείς επικισμούς. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν. σε ένα μεγάλο μέρος. Τώρα, τι άλλο μπορεί να γίνει σε σχέση με το σχέδιο του Τραμπ. Το σχέδιο αυτό είναι ένα είδος δημοψηφίσματος σε σχέση με το διεθνές δίκαιο τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, της δεκαετίες συνένωσης της κοινή πρωτεύουσα, της Ιερουσαλήμ, των επικισμών και ούτω καθεξής. Δηλαδή τι θέλει να κάνει αυτό το σχέδιο Τραμπ, Όλα, να, να οδηγήσει σε έναν εφησυχασμό. Δηλαδή να προσφύγει κανείς σε ένα δημοψήφισμα και να καταψηφίσει. Έχουμε διεθνείς παραμέτρους, το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας, θα πρέπει να αρκεστούμε σε αυτά, να βασιστούμε σε αυτά. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις, έτσι ώστε και άλλοι να καταψηφίσουν αυτό το σχέδιο. Επίσης, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να ε, σφυριλατήσει αυτό το σχέδιο Τραμπ. Και αυτές δεν είναι παραμερικές ιδέες, ένα σημείο εκκίνησης. Τώρα, το θέμα είναι κατά πόσο πραγματικά Πιστεύετε ή όχι στο διεθνές δίκαιο. Πιστεύετε στα δύο κράτη, ναι ή όχι. Αυτά βρίσκονται επιτάπητος και ελπίζω η απάντηση να να είναι θετική ως προς το διεθνές δίκαιο τα δύο κράτη και όχι ως προς τον συνεχή επικισμό και κατοχή. Ως προς το, την οργάνωσή μας δεν, δεν έχουμε σχέση με άλλους, ε, ε άλλους ε, ε, υπερασπιστές δημοσίου συμφέροντος. τώρα, σε σχέση με άλλες ΜΚΟ, όπως και άλλες ΜΚΟ, υπάρχει αυτή υπάρχουν αυτές οι ε, επιθέσεις κατά των μελών μας. Ε, για παράδειγμα, έγινε κλήτευση μελών μας από τον Ανώτατο Δικαστή γιατί δώσαμε ε, στοιχεία σε σχέση με στρατιώτες οι οποίοι μίλησαν κατά του ε, Ισραηλινού καθεστώτος. Γι' αυτό και έγινε και η κλήτευσή μας από τον ανώτατο δικαστή. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Έχουμε χρόνο και για έναν δεύτερο γύρο, εάν το επιθυμείτε. Ο κύριος Μπέρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαούλ. Ισχύει το ότι η οργάνωσή σας ε, στηρίζεται από απόστρατους ε, αλλά και εν ενεργεία στρατηγούς και στελέχη των μυστικών Έχετε τον λόγο. Νομίζω ε, ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ένα από τα βασικά στοιχεία εκείνης αυτής της εκστρατείας ήταν το, το εξής. Εγώ δεν ήθελα να ε, πάρω περισσότερο χρόνο του, ε, αλλά θα ήθελα να κατανοήσετε την εμβέλεια του όλου εγχειρήματος. Μιλάμε για ένα πολιτικό, πολιτικονομικό επίπεδο ε, δυστυχώς επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επιθέσεις, έλλειψη εμπιστοσύνης, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το νομικό σύστημα εναντίον μας. Θα ήθελα να σας δώσω μερικά παραδείγματα και μετά θα απαντήσω την ερώτηση, διότι έτσι αρμόζει καλύτερα τον Δεκέμβριο 15, Ιανουάριο του 16, 16 μέσα σε 16 εβδομάδες ε, υποστήκαμε πολλές επιθέσεις. Ε, τρεις φορές μας επιτέθηκε ο Νετανιάχου στην Ολομέλεια. Ο Υπουργός Εκπαίδευσης διέταξε να μην μας δέχονται τα σχολεία και πέρασε και τον νόμο κατά της οργανωσής μας. Ο Υπουργό Άμυνας έδωσε εντολή να μην μας δέχονται πουθενά σε κανένα σεμινάριο. Έγιναν ακροάσεις στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και ε, την Επιτροπή Ένομης Τάξης, όπου αναφέρθηκε ότι υπάρχουν ε, ανθρώπινες ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που στρέφονται κατά της ε, Ισραηλινής αρχής. Επίσης ε, έγινε ε, πρόταση από το κόμμα Λικούντ να απαγορεύσουν την δραστηριότητά μας. Επίσης, να μην είμαστε ούτε καν φεδρικοί στο στρατό, διότι υπηρετούμε άλλους αφέντες. Αυτό μέσα σε τρεις εβδομάδες και μόνο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μίλησα και ε, την κοινότητα η οποία έχει κλείσει στην Ιερουσαλήμ γιατί μας δέχτηκε. Επίσης στην Παρντεσράνα στο βορειοανατολικό Ισραήλ μας υποδέχτηκαν και μας άκουσαν και δυστυχώς η, το Ισραηλινό κράτος απαγόρευσε τη δραστηριότητα και κόβει τα κονδύλια αυτής της αρχής, αυτής της οργάνωσης. Αυτό το βλέπουμε και σε επίπεδο δημοτικών αρχών, όπου είχαμε και την υποστήριξη 330 πολιτών. Επίσης, στα περίχωρα του Τελαβίβ δώσαμε μία ε, συνέντευξη και εκεί πάλι απειλείται αυτή η οργάνωση και το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο απειλείται με περικοπή δαπανών. Και αυτό από το κόμμα του Λικούντ, το κόμμα του Νετανιάχου. Μας είχε καλέσει μία ε, βιβλιοθήκη και δυστυχώς τους υποχρέωσαν να σταματήσουν αυτή τη δραστηριότητα δεν τους ε, ενδιαφέρει αν πρόκειται για δραστηριότητες και ε, σεμινάρια, καθώς και διαλέξει υπέρ του Λικούντ. Μιλώ για μία πραγματικότητα όπου ε, ένα ζευγάρι σε ένα κιμπούτς στο βόρειο Ισραήλ, δύο αλίτες άρχισαν να τους επιτίθενται και αυτό το ζευγάρι είδε ένα άρθρο να δημοσιεύεται με τα ονόματά τους λέγοντας ότι καλέσαν, καλέσαν εκπροσώπους του, ε, ε, σπάζοντας τη σιωπή εμάς δηλαδή, και το κάναν επειδή δύο, οι δύο γη τους αυτοκτόνησαν ενώ υπηρετούσαν στο στρατό. Και τότε είχαμε την παρουσία 73 πολιτών. Μιλάω για μια πραγματικότητα όπου πρέπει να έχουμε φρουρούς έξω από τα γραφεία μας, διότι υποστήκαμε επιθέσεις. Κάποιος ε, συνελήφθη ο οποίος ε, ερχόταν προς τα γραφεία μας για να σου βάλει φωτιά. Και μπορώ να συνεχίσω στο διηνεκές. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δεν πρόκειται για λόγια. Και νομίζω ότι κάτι το ενθαρρυντικό είναι ότι βλέπουμε ανθρώπους που ποτέ πριν δημόσια δεν μας υποστήριξαν να το κάνουν πλέον. Κατανοώντας ότι αυτό ε, αφορά μία χώρα. Σε ποια χώρα θέλουμε να ζήσουμε και τι κάνει το Ισραήλ και η Ισραηλινή κοινωνία και πώς θέλει να ζήσει. Αυτό αφορά και την ε, Σαμπάκ η οποία όταν κλείσανε αυτή την, ε, αυτή την ε, καλλιτεχνική αίθουσα η οποία ήταν επρόκειτο να μας καλέσει είδαμε ότι δυστυχώς υπήρξε άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών και επίσης δημιουργήθηκε, οργανώθηκε μία διάλεξη ε, που φέρει τον τίτλο, έφερε τον τίτλο «Οι θεματοφύλακες σπάζουν τη σιωπή». Αυτό έγινε από, από μία από τις υπηρεσίες στρατού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι κάτι που βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο. Ιδιαίτερα στις υπηρεσίες ασφαλείας, πολλοί καταλαβαίνουν πού πάνε τα πράγματα και πού οδηγεί το Ισραήλ και η τρέχουσα κυβέρνηση και φοβούνται γι' αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και κάτι άλλο είναι πολλές δωρεές που δεχόμαστε από κοινού πολίτες. Έτσι συνδράμει ο μέσος Ισραηλινός θετικά και παίρνει και θέση. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ελπίζω εδώ να έχετε και εσείς το θάρρος να αντιταχθείτε, να μην δεχτείτε αυτή την πίεση, διότι έχει γίνει μεγάλος, μεγάλος πόλεμος, μεγάλη μάχη για την θεσμοθέτηση των ε, κατεχομένων που φτάνει και εδώ στην Ευρώπη, δηλαδή τι κατηγορίες ε, εκτοξεύονται από εκπροσώπους της Ισραηλινής κυβέρνησης εδώ στην Ευρώπη. Δηλαδή ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ θεωρείται και εναντίωση ή μάλλον εκδήλωση αντισημιτισμού και αυτή η εξίσωση είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να παίζουμε. Ο αντισημιτισμός είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να τον χειραγωγήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε ότι πολλοί εκπρόσωποι της κυβέρνησής μου κάνουν ακριβώς αυτό, το οποίο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας ευχαριστώ. Σαλίμα, έχετε κάτι ακόμα να πείτε και μετά θα δώσω τον λόγο στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο απέναντι σε όλα αυτά που ακούσαμε. Σίγουρα υπάρχουν μη καπάω μικρών παλαιστινιακέ ε, και ευχαριστώ την πρόεδρο που ανέφερε μία που ε, κάνουν αντίστοιχη προσπάθεια με τη δική σα και λένε όχι στη βία. Εσεί θα ήσασταν έτοιμοι να συνεργαστείτε με αυτές τις ε, ΜΚΟ μικρών και ίσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και φορείς θα είχαν ένα ρόλο για να υποστηριχθεί η άποψη των δύο κρατών του όχι στη βία της ε, πρωτεύουσα που μπορεί να είναι κοινή και για τους δύο νομίζω ότι υπάρχει εδώ πεδίο δράσης ή προσπάθειας. Θα έλεγα το εξή. Ε, αυτό το οποίο κάνει η οργάνωσή μας είναι ενημέρωση επίσης πολλές διαλέξεις, ε, συζητήσεις ε, σε σχολεία, πανεπιστήμια, ε, σε δημόσιους χώρους και περιοδίες. Στη Δυτική Όχθη 550 εκδηλώσεις το χρόνο, 13.000 άνθρωποι, κυρίως Ισραηλοί κάθε χρόνο μας ακούνε και Εβραίοι διεθνώς Οπότε όταν έρθετε στο Ισραήλ ευχαριστώ ε, να σας ε, συναντήσουμε, να σας δούμε με επιτόπου να σας δείξουμε τι συμβαίνει. Αλλά όταν πηγαίνουμε στην ε, Χευρώνα για να δούμε το τι συμβαίνει εκεί, ποια είναι η πραγματικότητα και ποιες είναι οι συνέπειες του επικισμού 850 επίκων ανάμεσα σε 200.000 Παλαιστινίους. Όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα που, έχουν, που έχει ο επικισμός. Ε, στην περιοχή Γάμα, εκτοπισμοί, κατεδαφίσεις σπιτιών. Όταν πηγαίνουμε στη Ραμάλα επίσης συναντάμε Παλαιστίνιους ακτιβιστές ε, και τις οικογένειές τους γιατί είναι σημαντικό για εμάς όταν έρχεται ο κόσμος εκεί να ακούει και την άλλη πλευρά και άλλη πλευρά. Δεν είναι η Ισραηλινή κυβέρνηση που είναι υπέρ της κατοχής ή η έπικη. Ε, κοιτάξτε, εγώ ήμουν στρατιώτης, ε, άσκησα την κατοχή με τα χέρια και τα πόδια μου. Οι άλλοι είναι αυτοί που την υφίστανται όμως. Αυτή είναι η άλλη πλευρά, η Παλαιστίνη. Και εκεί πέρα συναντάει ο κόσμος και την άλλη πλευρά και τους μιλάει. Σημαντικό αυτό για τους νεαρούς ε, Ισραηλινούς στα σχολεία και στα στρατιωτικά σχολεία. Πολλούς από αυτούς είναι η πρώτη φορά στη ζωή τους που συναντάνε Παλαιστίνιο και μπαίνουν σε σπίτι Παλαιστίνιο. Και ακούνε τους Παλαιστινίους να τους μιλάνε και έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω πόσο σημαντικό είναι ο σεβασμό ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και της ελευθερίας σε μια περιοχή όπου υπάρχει σύγκρουση τα τελευταία 70 χρόνια. Χτες το βράδυ επέστρεψα από εκεί. Μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα έχουμε αιτήσιες συναντήσεις και με τις δύο πλευρές, Ισραηλινούς, Παλαιστίνιους και αυτό το οποίο μπορούμε να επιβεβαιάσουμε είναι αυτό το οποίο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι πως οπωσδήποτε μειώνεται ο χώρος τη κοινωνίας των πολιτών στο Ισραήλ αλλά και στην Παλαιστινιακή κοινωνία. Μας ανησυχεί ιδιαίτερω η δυνατότητα τη κοινωνίας των πολιτών και ειδικά των υπερασπιστών ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις δύο πλευρές. Και αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Σαούλ οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται κατά τις οργάνωσης αυτής και άλλων επίσης ε, έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν λήψεις και από την Παλαιστινιακή πλευρά και δεν θέλω καν να αναφερθώ στην Χαμάς ε, μια τρομοκρατική οργάνωση κτλ. Και την Ισλαμική Τζιχάτ και τα σχετικά είναι και αυτό το οποίο πρέπει να δούμε. Κάποιος ε, το ανέφερε να ακουστούν και οι δύο πλευρέ. αλλά αυτό το οποίο κάνουμε στις πολιτικές επαφέ μας με τις δύο πλευρές τονίζουμε όλο και περισσότερο την σημασία της κοινωνίας των πολιτών, ε, των υπερασπισμών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις δύο πλευρές. Για εμάς λοιπόν αυτό είναι ένα στοιχείο ειρηνευτικό, γιατί όποιο σχέδιο και αν υπάρξει κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει δεκτό από τους ανθρώπους, όχι μόνο από τους πολιτικούς ε, και τις ε, κυβερνήσεις. Όταν υπάρχει το πιο τέλειο σχέδιο. Αν η κοινωνία των πολιτών δεν το δέχεται, ε, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να το δεχτούν οι πολίτες και των δύο χωρών. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια είναι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών και στις δύο πλευρές. Κομισιόν σχετικά προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσπαθούμε να αυξήσουμε και τη χρηματοδότηση οπότε προφανώς μία ΜΚΟ όπως η Σπάζοντας την Σιωπή με βάση τις ε, δραστηριότητες της ε, έχει μεγάλη σημασία και είναι σημαντικό να διατηρηθεί η κοινωνία των πολιτών. Τελευταία παρατήρηση. Πολλές φορές ε, συναντιέμαι με εκπροσώπους των ΜΚΙΟ και όλο και πιο συχνά από την Παλαιστινιακή πλευρά μας λένε «Κοιτάξτε, θέλετε να συζητήσουμε με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μιας χώρας που έχει πάρει τη γη μας, ε, σκοτώνει τους δικούς μας. Ε, πώς θα γίνει αυτό. Το λέω γιατί έχουμε όλο και περισσότερα προβλήματα για να αναπτύξουμε κοινά προγράμματα μεταξύ των ΜΚΟ της κάθε πλευράς. Γιατί υπάρχει άρνηση ναι, για να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι και αυτό κάτι το οποίο εξετάζουμε ε, αυτή τη στιγμή. Και συνοψίζοντας ε, και θέλουμε την στήριξή σας θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενίσχυση της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών και στις δύο πλευρές. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, Γεχούντα. Και υπόσχομαι ότι οπωσδήποτε θα έρθουμε να μας τα πείτε εκεί πέρα. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στην επόμενη συζήτηση. Um, θα ζητούσα από όλους. Voilà. Donc je vais, on va commencer le sixième point. Να πάμε λοιπόν ε, στο σημείο 6. Αν θέλετε να καθίσετε θα είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, όπως τα γνωρίζετε, το σημείο 6 Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα σε όλα τα θέματα. Εδώ μιλούμε για το σεβασμό των ε, μειονοτήτων, των ε, πεπιθήσεων και των ε, θρησκειών. Της θρησκευτική πίστης. Λοιπόν, οι τελευταίες δημογραφικές και εγγραφικές μελέτες δείχνουν ταχύτατες αλλαγές που επηρεάζουν τις τη θρησκευτική και τη φιλοσοφική πίστη σε παγκοσμία κλίμακα και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε επίσης ε, μια αύξηση της ποικιλότητα ε, νέων μορφών πνευματικότητας και χαρισματικών κινημάτων, λέει η Πρόεδρος. Δυστυχώς παρατηρούμε επίσης και την άνοδο του φονταμεταλισμού και του εξτρεμισμού στα θρησκευτικά πλαίσια. Θα περιμένω λίγο να βγείτε, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επαναβεβαιώνουμε την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκευτικής πίστης ε, είναι βασικές αρχές και έννοιες της δημοκρατικής μας ε, κοινωνίας και κατά των καταχρήσεων. Ε, βλέπουμε, σημειώνουμε παντού στον κόσμο παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών και διωγμούς ενεργητικές διακρίσεις κατά πολιτών, ανθρώπων που έχουν κάποια άλλη πεποίθηση ή θρησκεία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικοί, να μην έχουμε διακρίσεις και αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε σήμερα το απόγευμα ε, για τον αντίκτυπο και το αποτύπωμα, το παγκόσμιο της συνύπαρξης των θρησκειών αυτών και για τις ε, καλύτερες πρακτικές που μπορούμε να έχουμε για να διαχειριστούμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω τον κύριο Έριν Βίλσον, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χρόνιγκεν στην Ολλανδία. Τον κύριο Μουχαμάντ Νουρντίν Λεμού, καθηγητή έρευνας ε, στο Ίδρυμα Ντάουα στην Νιγηρία για, την, ε, για τον διάλογο μεταξύ των δογμάτων των θρησκευτικών στη χώρα του, την κυρία Σιμάνσκι που είναι επικεφαλής ε, του Ιδρύματος ε, της ε, Καθολικής Εκκλησίας σε μπάση περιπτώσει ε, ας ξεκινήσουμε με την κυρία Βίλσον. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα. Ε, καλό απόγευμα Πρόεδρε, αγαπητά αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Μιλούμε για ένα παγκόσμιο δικαίωμα που είναι εξίσου σημαντικό όπως και τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έχουμε ιδιαιτερότητες στην προστασία του οι οποίε έχουν επιπτώσει για το σεβασμό των μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια και περιβάλλοντα. Θα εστιαστώ σε τρει τέτοιε προκλήσει για την καλύτερη κατανόηση της θρησκεία και των δικαιωμάτων. Αυτά προκύπτουν από πρόσφατε έρευνε, επί μελέτες μάλλον που έγιναν επί του θέματο αυτού, όπου κάναμε ε, μαζί με συναδέλφους του ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου στην Ινδονησία και στην Ινδία. Πρώτον, πώς πρέπει να κατανοεί κανεί να αντιλαμβάνεται τη θρησκεία και την πεποίθηση. Οι αναλυτές, οι ακαδημαϊκοί του θέματος λένε αφενός ότι μπορεί να μην έχουμε έναν συνολικό παγκόσμιο ορισμό της θρησκείας, αλλά αναγνωρίζουμε τι είναι όταν το βλέπουμε. Αυτή η κοινή κατανόηση, η ερμηνεία, ε, προϋποθέτει ένα κοινό ιστορικό, μια κοινή ιστορική παράδοση η οποία δεν υφίσταται πάντα. Και ακριβώς η αντίθεση του να φτάσουμε σε έναν ε, παγκόσμια συμπεφωνημένο ορισμό της θρησκείας δείχνουν οι επικριτές της θέσης αυτής και τονίζουν ότι η θρησκεία είναι ένα ρευστό, πολύ σύγχρονο νόημα Η Πρόεδρος ε, ευτυχώς ε, διακόπτει την ομιλήτρια για να τη ζητήσει να μιλάει λίγο πιο αργά. Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο. Ως προς την ανάδειξη λοιπόν κοσμικών αντιλήψεων που δείχνουν ότι η θρησκεία είναι κάτι που πρέπει να το διακρίνουμε απολύτως από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αμφισημία για το πώς διακρίνουμε πεποίθηση ή θρησκεία είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση των μειονοτικών πληθυσμών. Οι κυβερνήσεις έτσι μπορούν να αποφασίζουν ποιες πεπιθήσεις ή τάσεις ή έθιμα δεν είναι θρησκεία και επομένως δεν προστατεύονται από τον νόμο. Χρησιμοποιείται Επίσης, καμία φορά ε, καταβάλλονται προσπάθειες για την προστασία των ομάδων αυτών που καταλήγουν σε περισσότερες αρνητικές παρά θετικές συνέπειες. Γιατί συχνά στοχοποιούνται και υφίστανται ακόμα πιο έντονε διακρίσεις. Η έρευνά μας στο Κουτζαράτ έδειξε ότι το δικαίωμα στο οποίο προσδοκούσαν οι, τα μέλη της μειονοτικής εκεί κοινότητας ήταν το δικαίωμά τους στην, όχι στο να διαδηλώνουν την πεποίθησή τους, αλλά στο να μην υφίσταται διακρίσεις. Έχουμε πολλά παραδείγματα όπως οι κόπτες στην Αίγυπτο μεταξύ άλλων, αλλά εν πάση περιπτώσει η παραβίαση των δικαιωμάτων επί τη βάση της θρησκευτική ταυτότητας ίσως να μην είναι η πιο αποτελεσματική διόδοση της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Άλλη μια πρόκληση είναι η γλώσσα και η αμφισβήτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κοινωνικό και ιστορικό οικοδόμημα της ούτως αποκαλούμενης δύσεως. Λένε πολλοί ότι αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η έννοια αυτή, προκύπτουν από την παράδοση του δυτικού αφηγήματο. Η διαφωνία σχετικά με την προέλευση, την αρχική προέλευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιείται και στον πολιτικό λόγο, ώστε να αρνηθεί κανείς συγκεκριμένα δικαιώματα σε συγκεκριμένες ομάδες ή χώρες, δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΔ, της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας πίστης. Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ελευθερία έκφρασης και ε, πεποίθησης μάλλον και πίστης σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού οι γυναίκες και οι ΛΟΑΔ έχουν και αυτή δικαίωμα ανεξιθρησκείας, δικαίωμα ελευθερίας πίστης. Ο διάλογος αυτός για την προέλευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιπτώσει στην πράξη, προσπαθώντας να πείσει τους ε, ανθρώπους για το ένα ή το άλλο και συνήθως είναι μια μάταιη προσπάθεια. Υπό μία έννοια δεν έχει καμία σημασία αν μπορούμε να αποδείξουμε την προέλευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϊόν του δυτικού πολιτισμού ή πολλαπλών πολιτισμών. Οι διαφωνίες που υφίστανται υφίστανται για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Πιο ρεαλιστικά θα έπρεπε κανείς να αναγνωρίζει, να γνωρίζει καλύτερα την διαφορετική ανάγκη πίστης και έκφρασης σε διάφορες κοινωνίες και χώρες. Στην Αίγυπτο, στην Κίνα, στην Ινδονησία, στην Ουγγάντα, για να δώσουμε μόνο λίγα παράδειγμα, λίγα παραδείγματα, η προστασία της αξιοπρέπειας και της ισότητας περνάει μέσα από την προστασία της ανεξιθρησκείας και της πεποίθησης. Οι αρχές που ενέχονται όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν απήχηση σε διάφορες γλώσσες και σε διάφορες παραδόσεις. Πρέπει να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις, να εστιαζόμαστε στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας ή της κάθε κοινωνίας όταν αναπτύσσουμε ε, σχέδια ή πλαίσια προσιλοποίηση. Τώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ ατομικών και κοινοτικών δικαιωμάτων. Στα πλαίσια της ανεξιθρησκείας αυτό επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο διότι έρχεται να προσθεθεί η έννοια της θρησκείας ή της πίστης η οποία πολύ συχνά γίνεται αντιληπτή εσωτερικά ως δικαίωμα του κάθε ατόμου να πιστεύει σε ένα πλαίσιο αρχών ή αξιών ή ενιών. Όμως αυτή η ερμηνεία που είναι αρκετά δυτικόστροφη ή προτεσταντική, για να το πούμε έτσι, δεν είναι ευκόλως κατανοητή στην Ινδία, για παράδειγμα, όπου η θρησκεία είναι αντιληπτή, γίνεται αντιληπτή ως ίδιων μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας, μιας εθνικής ομάδας, μιας κοινωνικής ομάδας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ένα άτομο μπορεί να έχει πολλαπλές θρησκευτικέ ε, ε, τάσεις, δηλαδή να είναι πολιτιστικά μουσουλμάνος κανείς, ενώ στην πράξη να είναι άθεος ή και χριστιανός. Αυτά έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την ανεξιθρησκεία και την πεποίθηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το δικαίωμα αυτό αναφέρεται ως δικαίωμα της ανεξιθρησκείας στον Καναδά, στις ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγαλύτερη προσοχή ως δικαίωμα στην πίστη. Ελευθερία θρησκευτικής πίστης. Και πολύ συχνά υπάρχει μια επίκριση ότι υπάρχει μια επιμόλυνση από χριστιανικές ιδέες ή παραδόσεις των ενιών αυτών. Οι διακρίσεις αυτές είναι λιγότερο σημαντικές σε ένα ευρύτερο ε, πλαίσιο και σε μια ευρύτερη παγκόσμια συζήτηση. Είτε μιλούμε για φόρμα από τα αρχικά της ελευθερίας πίστης και πεποίθησης, είτε για ανοιξή θρησκεία, είναι σημαντικό να δούμε ότι εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερων ε, πρωτοβουλειών πολιτικής για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού ή της τρομοκρατίας, ε, βίαιων ενεργειών, βίαιων ομάδων. Πολύ συχνά περι, χρησιμοποιούμε τέτοια φαινόμενα, βία φαινόμενα ή την καταπολέμησή τους προκειμένου να περιορίσουμε την ελευθερία στη θρησκεία ή στην πεποίθηση. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε ε, χώρες ε, πλειοψηφικά μουσουλμανικές. Για το πώς ε, βλέπουν δηλαδή με καχυποψία τις ελεύθερες θρησκευτικέ πεπιθήσεις συγκεκριμένες κυβερνήσεις ή ηγεσίε των χωρών αυτών. Και αυτό προεκτείνεται και σε πολιτισμικά ήθη και έθιμα όπως η χρήση ή όχι ε, του καλύματος της κεφαλής από τις γυναίκες. Είναι η γλώσσα πάντως της ελευθερίας θρησκείας και πεποίθησης και όχι η αντίσταση στο ίδιο το δικαίωμα που δίνει ουσία στη μελέτη που κάναμε και στις δύο περιοχές στην Ινδία και στην Ινδονησία. Χρησιμοποίησαμε προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τοπική γλώσσα ώστε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων δίνοντας έμφαση όχι στις διαφορές μεταξύ τους, αλλά σε κοινά προβλήματα, κοινέ προκλήσεις, πώς μπορούν από κοινού να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που υφίσταται για τους δύο ή για τις περισσότερες κοινότητες η κατανόηση των διαφορών με την άλλη κοινότητα βοηθά σε μια οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Η ελευθερία πίστης έχει διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με το που βρισκόμαστε, ανάλογα με το αν ο λόγος αυτής της ανεξιθρησκεία ή ελευθερίας πίστης πρέπει να αξιολογηθεί προς το πολιτισμικό, περιβαλλοντικό ή οικονομικό πλαίσιο και τους φορείς που ε, ενεργοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά σε όλα τα πλαίσια οι βασικές αρχές και έννοιες της ελευθερίας πίστης υφίστανται παντού. Σεβασμός για άλλες θρησκευτικές πεπιθήσεις, ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμός για όλους τους ανθρώπους. Το ερώτημα του πώς καθορίζει κανείς τη θρησκεία με τις διαφορετικές ερμηνείες της και αποχρώσεις της είναι σημαντικό για τους ακαδημαϊκούς, όχι αναγκαστικά όμως για τους ηθήνοντες ε, της πολιτικής. Ε, όταν μιλούμε για την προστασία της ανεξιθρησκείας, οι ίδιοι οι πολιτικοί υπεύθυνοι αρμόδιοι ε, καλούνται ενεργά πρακτικά να ορίσουν την ανεξιθρησκεία ή τη θρησκευτική πίστη χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται. μιλούμε για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των μειονοτικών πληθυσμών που είναι το πιο σημαντικό για τους υπευθύνου. Σα ευχαριστώ λέει πρόεδρο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μουχαμάτ Νουρουντίν. Έχει το λόγο για 10 λεπτά επίση περίπου. Good afternoon and... Καλησπέρα σας ε, και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εγώ θα ήθελα να εξετάσω στρατηγικές ε, διαλόγου μεταξύ των θρησκειών ε, για να στηρίξουμε την ανεξιθρησκεία. και τέτοιες ε, κοινωνίες. Θα ξεκινήσω με μία δήλωση του Αμπουχαμίντ Αλγκαζάλη, ενός μουσουλμάνου νομικού, που είπε «Οι φίλοι είναι τεσσάρων ειδών. Κάποιοι είναι σαν το φαγητό ωφελείουν και τους χρειάζεσαι. Κάποιοι άλλοι φίλοι είναι σαν το φάρμακο. Δεν τους χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν έχεις δυσκολίες τους χρειάζεσαι. Κάποιοι άλλοι φίλοι είναι σαν την αρρώστια. Σε εξασθενούν και σε κάνουν λιγότερο παραγωγικό. Και το τέταρτο είδος είναι σαν δηλητήριο, σε σκοτώνουν. Όταν μιλάμε για τις σχέσεις μας ε, μεταξύ των κοινοτήτων και εντός των ε, κοινοτήτων και το πώς βλέπουμε τον ε, διαθρησκευτικό διάλογο και πώς βλέπουν την ανοιξή θρησκεία, παρατηρούμε ότι υπάρχουν μέλη κάθε κοινότητας που θέλουν να οικοδομήσουν γέφυρες. Το θεωρούν θετικό με βάση κάποια πιστεύω τους. Άλλοι λένε ότι αν μας βολεύει να το κάνουμε. Αν δεν μας βολεύει, όχι από μόνο του, αλλά αν είναι καλό. Άλλοι ε, θα το ανεχτούν, αλλά δεν, ε, το, δεν τρελαίνονται κιόλα. Άλλοι θεωρούν ότι υπονομεύει την ταυτότητά τους. Είναι δύσκολο λοιπόν να πούμε ότι η τάδε κοινότητα ε, θέλει ή δεν θέλει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις γενικεύσεις. Ο παραδοσιακός κανόνας ε, του θρησκευτικού διαλόγου είναι ας πούμε η οικοδόμηση γεφυρών και μια άτυπη ε, συνθήκη ειρήνης θα λέγαμε. Και αυτό περιλαμβάνει τις μεγάλες ε, θρησκείες, δηλαδή στην Ιγυρία μουσουλμάνοι χριστιανοί. Το κλίμα όμως αλλάζει. οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Έχουμε διαφορετικές ε, πτυχές ε, της άκρας ε, δεξιάς εθνικιστικών, φονταμενταλιστικών, ακραίων κινημάτων. Όλα αυτά τροφοδοτούν το ένα το άλλο. μία πλευρά προκαλεί και προκαλεί την άλλη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε τώρα στο πλαίσιο αυτό όταν ε, θέλουμε να κοιτάξουμε το πώς ο διαθρησκευτικός διάλογος μπορεί να προωθήσει την ε, άνεξη θρησκεία, βλέπουμε ότι υπάρχουν νέοι παίκτες και νέα ζητήματα. Δυστυχώς ε, σε πολλές κοινωνίες ο διασκευτικός διάλογος, δηλαδή εάν δω την Νιγηρία, δεν έχει γίνει τίποτα περισσότερο από μια γέφυρα. Δηλαδή οι ηγέτε δεν πλακώνονται. Αλλά δεν εκπροσωπούν ε, τη μάζα. Οι ηγέτε είναι elite. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε 100 άτομα στην Ιγυρία και δεν θα τους ακούσει το Άισις. Μπορούν η Σαουδική Αραβία να βρουν 100 διανοούμενους, δεν θα τους ακούσει το Άισις. Δηλαδή οι άνθρωποι στην βάση δεν ακούν αυτούς που υποτίθεται ότι τους εκπροσωπούν στον διαθρησκευτικό διάλογο. Όπως είπαμε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αισθάνονται και αναγκάζονται να αναγνωρίσουν ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης ε, ε, είσαι πλειοψηφία στον τόπο σου, αλλά θα υπάρχουν πάντα μειονότητε ε, παντού. Και αν ε, είναι να υπάρχει αμοιβαιότητα και θέλεις ε, θρησκευτική ελευθερία για τη δική σου τη μειονότητα, πρέπει να υπάρχει ανεξιθρησκεία και για τις μειονότητες στο δικό στον τόπο. Οπότε είναι ο χρυσό κανόνας, να μην κάνει αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Για άλλου βεβαίω. Το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν θέμε άλλους πολέμους, οπότε θα πρέπει να υπερισχύσει α, το ευρύτερο καλό, το κοινό καλό. Ο διασκευτικός διάλογος συνήθως ξεκινά με τη λεγόμενη αρμονία και μετά περνάμε στα ε, κοινωνικά ζητήματα. Όπως είπα, συχνά δεν πάμε παραπέρα από αυτό. Οπότε το να αναμένουμε ο διαθρησκευτικός διάλογος να αρχίσει να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα είναι δύσκολο. Καλό να δούμε τι μπορεί να κάνει ο, ο ενδοθρησκευτικός διάλογος. Τι μπορούν να κάνουν οι δηλαδή και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λέω ότι είναι άχρηστος, αλλά λέω ότι για καλύτερα αποτελέσματα το καλύτερο είναι ο ενδοθρησκευτικός διάλογος και θα επανέλθω σε αυτό. Όμως, για να έχουμε διαθρησκευτικό διάλογο χρειάζεται καλύτερη οικοδόμηση γεφυρών. Ε, πραγματικών γεφυρών. Δηλαδή, ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφορά τις κοινότητες, όχι μια γέφυρα στο πουθενά που δεν αφορά κανέναν. Πρέπει να είναι εντός της κοινότητας αυτής. Αλλιώς θα έχουμε ακριβώς τους ηγέτες ε, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τα στερεότυπα αυτά. Γιατί βεβαίω όταν έρχομαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους ε, συνήθως πηγαίνουμε κατευθείαν στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και οι θρησκευτικοί ηγέτες οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα διαχείρισης συγκρούσεων κτλ. Ε, προσπαθούν ακριβώς να περάσουν την εκπαίδευση αυτή ε, εκεί όπου χρειάζεται γιατί οι ηγέτες δεν εμπλέκονται στα πραγματικά προβλήματα και καμιά φορά βλέπουμε όλα αυτά τα ζητήματα δηλαδή οι ηγέτες πηγαίνουν ξανά και ξανά εκεί πέρα στα σεμινάρια αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφείς ε, προσδοκίες για τα αποτελέσματα του διασκευτικού διαλόγου. Αλλιώς έχουμε μεγάλες προσδοκίες και πενιχρά αποτελέσματα. Δηλαδή θεωρούν ότι ο διάλογος αυτός είναι αντιβιωτικό ευρέως φάσματος που κάνει τα πάντα που θα λύσει όλα τα προβλήματα, ενώ τα προβλήματα καμιά φορά δεν σχετίζονται με την θρησκεία. Για να λειτουργήσει λοιπόν ο διάλογος αυτός θα πρέπει κάθε πλευρά να έχει στέρεες βάσεις. Δεν μπορεί να χτίσουμε μια σοβαρή γέφυρα χωρίς σωστά θεμέλια. Η γέφυρα δεν πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει σε κάποιον άλλον. Ε, είναι μια γέφυρα μεταξύ των δύο αλλά δεν ανήκει σε μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει όσοι συμμετέχουν στον ε, διάλογο να αναγνωριστούν ως ε, πραγματικοί εκπρόσωποι των κοινοτήτων. Γι' αυτό ακριβώς ε, βλέπουμε ότι είναι διάφοροι έτοιμοι να μιλήσουν, αλλά οι κοινότητες δεν τους ακολουθούν. λένε πήγαινε εσύ μίλα, εμείς ε, έχουμε τη δική μας πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν όταν οικοδομείς μία γέφυρα να μην ξεκινάς από τη μία πλευρά και φτάνει στην άλλη, ε, η γέφυρα ξεκινά και από τις δύο πλεύρε να χτίζεται. Και βεβαίω οικοδομείται με βάση την εμπιστοσύνη. Όσο περισσότερη εμπιστοσύνη υπάρχει, τόσο πιο σοβαρά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν, αν θέλετε. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την οικοδόμηση γεφυρών θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κοινότητες πραγματικά θα θεωρήσουν αυτή τη γέφυρα δική τους. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να την προστατεύσουν και να μην αφήσουν άλλους να την κάψουν. Αυτοί οι οποίοι καίνε τις γέφυρες δεν μπορεί να είναι η πινελόπη ε, το πρωί να πλέκει και το βράδυ να ξεπλέκει. Δεν προκειμένου δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι το βράδυ ε, στα κοινωνικά μέσα να υπονομεύουν ε, τις προσπάθειες. Όσον αφορά την ταυτοποίηση των προβλημάτων, ε, θα αναφερθώ πάλι στην Ιγυρία που γνωρίζω. Μια μεγάλη χώρα, τεράστια, και για να χρησιμοποιήσω μια μεταφορά, η Ιγυρία έχει πολλές λακκούβες στους δρόμους της. Οι λακκούβες υπάρχουν σε όλες τις χώρες, δεν έχω δει εδώ ακόμα αλλά παρόμοιε είναι. Την ίδια ζημιά κάνουν. Αλλά επειδή είναι παρόμοιε. δεν σημαίνει ότι έχουν παντού τις ίδιες αιτίε ή τις ίδιες λύσεις. Μπορεί να προκαλούνται από ε, κακή ποιότητα. ποιότητας. Ε, μπορεί να προκαλούνται από τον παγετό ή από την υπερβολική ζέστη. Ε, μπορεί να είναι βαρέα οχήματα. Μπορεί να είναι κακή κατασκευή, κακή άσφαλτος. Είναι ένα συνδυασμό διαφόρων πραγμάτων. Όταν λοιπόν μιλάμε για ζητήματα που σχετίζονται με τον διαθυσκευτικό ε, διάλογο πρέπει να σκεφτόμαστε και να δρούμε τοπικά. Καλό είναι να δούμε το τι γίνεται αλλού, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι για εμάς χωρίς εμάς. Ε, δεν μπορεί να γίνει κάτι για την τοπική κοινότητα χωρίς συμμετοχή της. Αν προσπαθήσουμε να πάμε πάρα πολύ γρήγορα με μία ε, ύπεθρο της κοινότητας αυτής. Λένε ε, για να πας μακριά χρειάζεσαι και άλλους. Για να πας γρήγορα μόνο. μόνος Λοιπόν, δεν θα πρέπει να έχουμε διάφορα στερεότυπα όπως έχουμε δει παραδείγματο χάρη στον Ταρφούρ και αλλού όπου ήρθε ο κόσμος με τις δικές του προκαταλήψει, τους έδωσαν διαβεβαιώσεις θεώρησαν ότι βρέθηκε μια λύση αλλά δυστυχώ δεν άγγιξαν τι αιτίε. οπότε για να προσπαθήσουμε πραγματικά να βρούμε τον ρόλο της θρησκείας σε οποιοδήποτε στιγμή. Είτε μιλάμε για ανεξιθρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Όταν βρούμε και πούμε ότι ένα ζήτημα σχετίζεται με τη θρησκεία, πρέπει να θυμόμαστε ότι η θρησκευτική μεταρρύθμιση δεν είναι ποτέ κάτι το οποίο έρχεται από τα έξω. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι καθολικός να κάνει την καθολική εκκλησία να αλλάξει. Ούτε τους μουσουλμάνους. Πρέπει αυτοί που είναι μέσα να συμφωνήσουν ότι πρέπει να αλλάξουμε τη θέση μας σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να ε, δούμε με ποιον μιλάμε, σε ποιον δίνουμε πληροφορίες. Μπορεί να αφορά τον ε, γενετήσιο ακροτηριασμό ή ένα αφήγημα που προωθούν κάποιοι ή τους νόμους περί βλασιμίας, οτιδήποτε και αν είναι. Περισσότεροι ηγέτες ε, είναι λίγο όπου φυσάει ο άνεμος. Είναι σαν τις σημαίες. Αλλά η σημαία δεν καθορίζει το από που φυσάει ο άνεμος. Α, αρκετοί ηγέτες ε, κοιτάνε προς τα που φυσάει ο άνεμος και μετά εκδηλώνονται. Ελάχιστοι μπορούν να επηρεάσουν την κατεύθυνση στην οποία φυσάει ο άνεμος και έχουν αρκετές επαφές για να αλλάξουν το τι πορεία ακολουθεί η κοινότητά τους. Άρα είναι σημαντικό να μπορούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε τα κλειδιά και είναι οι φύλακες του γαλαξία του θρησκευτικού γαλαξία. Οι θρησκείε εξελίσσονται, επηρεάζονται από τον πολιτισμό και από διάφορα πράγματα και στο μουσουλμανικό περιβάλλον υπάρχουν ε, οι μουφτίδες, ε, οι ειδικοί. Δεν είναι απλά διανοούμενοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια εσωτερική μεταρρύθμιση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σεβαστοί αλλά συνήθως είναι άγνωστη στην πλειοψηφία. Οπότε αν θέλουμε να αλλάξουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ε, σημαντικό είναι να δούμε εάν μας ακούνε αυτοί οι συγκεκριμένοι λόγοι. Εάν το πιστέψουν, το κάνουν δικό τους και δεν το... Δεν λένε ότι κάποιος άλλος θέλει να κάνουμε αυτό, λένε όχι, πρέπει να αλλάξουμε θέση, γιατί ε, έχουμε τα εξή ωφέλη ας πούμε ή γιατί θα χάσουμε εάν δεν αλλάξουμε. Και μόλις βρούμε αυτήν την ομάδα και μοιραστούμε τις πληροφορίες και το θεωρήσουν κάτι δικό τους, μετά κοιτάνε ποιος θα είναι ο επόμενος. Είναι η πανεπιστημιακοί. Τότε έρχονται οι πιο χαρισματικοί ηγέτες και όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία αρχίζει να φυσάει ο άνεμος και τότε οι ηγέτες των διαφόρων ε, κοινοτήτων που σε πολλές ε, περιπτώσεις θέλουν να ξέρουν προς τα που ψάει τότε αναλαμβάνουν. Το είδαμε αυτό όταν προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της πολιομιελίτιδας στην Ιγυρία. Κάποιοι λέγανε ότι το εμβόλιο στηρώνει τον πληθυσμό. Ε, κυκλοφών διάφορες συνωμοσίες. Ε, όταν λοιπόν οι λόγοι ήρθαν σε επαφή με τους ειδικού και τα σχετικά άρχισαν να εκπαιδεύουν και άλλους ε, και άρχισε ε, το θέμα να φτάνει στη βάση και μέχρι τότε ε, ήταν εύκολο οι πολιτικοί ηγέτες να νομοθετήσουν χωρίς καμία αντίσταση. Θα σταματήσω εδώ και θα πω απλά πως υπάρχει ανάγκη να κινούμαστε προσεκτικά όταν θέλουμε να αλλάξουν ε, θρησκευτικές θέσεις αν δεν υπάρχει η συμμετοχή ακριβώς των θεματοφυλάκων του θρησκευτικού αφηγήματο. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στη Μαρτσέλα Ζημάνσκι. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για αυτά τα 10 λεπτά που μου δίνετε για σας πω ότι με απασχολεί από το 2003 και μετά. Ήμουν ε, επικεφαλής ε, λόμπι και τότε ασχολήθηκα πρωτίστως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασχολήθηκα στη χώρα μου στο Μεξικό μετά από την εξέγερση των Σαπατίστας. Όπως ξέρετε, ε, μετά ε, ελήφθησαν υπόψη θετικά μέτρα και οι αυτόχρονες ε, πληθυσμοί μπόρεσαν να ορίσουν ε, ένα σύνορο για να μπορέσουν να δράσουν. Η Μαρία ήθελε να σπουδάσει δημοσιογράφος και όμως στην κοινότητά της ε, δεν επιτρεπόταν η εκπαίδευση στις γυναίκες. Δεν, δεν μπόρεσε λοιπόν να ε, μεταβεί πέρα από τα σύνορα, διότι οι πρεσβύτεροι του χωριού της είπαν όχι. Έτσι, ως άνθρωπος και ως Μεξικανή δεν μπόρεσε να ε, εκπαιδευτεί, δεν μπορούσε να έχει λόγο και άλλοι Μεξικανοί είτε στο εξωτερικό είτε στο Μεξικό δεν μπόρεσαν να την υπερασπιστούν. Όλα αυτά με εξέπληξαν. Η Μαρία ήθελε να είναι ελεύθερη και να ακολουθήσει τη συνείδησή της και αυτό που ήθελε να σπουδάσει. Και θεώρησε ότι είναι ίση με τις κοπέλες στο διπλανό χωριό. Όμως δεν ήταν τα καθολικά δικαιώματα, δεν ίσχυαν για εκείνη. Δεν μπορούσε πλέον να αποφασίσει πώς θα σκεφτεί και δεν μπορούσε να ζήσει τη ζωή της όπως ήθελε. Αυτά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, δυνάμει του άρθρου 18 της ε, θεμελιώδους ε, δήλωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορά την αναζήτηση της αλήθειας, να μπορέσει κανείς να δεχτεί παγκόσμιες αρχές. Δυστυχώς όμως ε, τα ανθρώπινα όντα δεν το επιτρέπουν. Η Μαρία είναι ένα από τα παραδείγματα, αλλά θα μπορούσαμε να επεκταθούμε σε ευρύτερη κλίμακα για να μην δεχτούμε την ε, ποικιλότητα και την πολυπικιλότητα της ε, σκέψης ε, δείτε την περίπτωση της Κίνας και της ε, τεχνητής νοημοσύνης. 500 εκατομμύρια κάμερες μπορούν να παρακολουθήσουν τα δύο δις ε, κατοίκους. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνδράμει και η οργάνωση της οποίας ηγούμε η Εκκλησία σε κίνδυνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε. Δύναμη του άρθρου 18 που, έχει, που είναι ύψης της σημασίας και για τις ε, εμπόλεμες και στις εμπόλεμες ζώνες. Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι είναι, ε, φέρουν αξιοπρέπεια, είναι ίσοι ενώπιον του Θεού και αυτό θα πρέπει να ισχύει σε κάθε επίπεδο. Σε επίπεδο κρατικό, ε, θρησκευτικό, διαθρησκευτικό και ούτω καθεξής. Στις εμπόλεμες ζώνες βλέπει η Εκκλησία πώς οι άνθρωποι χάνουν την ελευθερία τους, πεθαίνουν και η ε, ελεύθερη συνείδηση είναι και το τελευταίο κομμάτι. Έχουμε μία ετήσια, ε, μάλλον ε, διετή έκθαση, την, η οποία έχει 180 σελίδες και μιλάμε για ε, την εφαρμογή του άρθρου 18 εκτός είπα και αυτό αφορά 196 χώρες και τις βασικές θρησκείες. Δημοσιεύεται σε έξι γλώσσες και μπορείτε να το ε, συμβουλευτείτε και διαδικτυακά. Η επόμενη έκδοση προβλέπεται για τον Οκτώβριο του 2020. Ασχολούμε πυρετοδός με αυτήν η έκδοση αυτή ε, δεν ε, εκδίδεται από μια κυβέρνηση, απλώς θέλει να συνδράμει το κοινό και τους ε, πολιτικούς, αυτούς που καθορίζουν πολιτικές. Ανέφερα τη Μαρία, διότι στην ουσία συρρυκνώνονται τα δικαιώματά της επειδή το αποφασίσουν κάποιοι άλλοι. Θα πρέπει εμείς να συνδράμουμε ώστε να μπορέσει κανείς να δράσει όπως επιθυμεί, να μην καταπατώνται, με συγχωρείτε, τα ανθρώπινα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να ε, κατατροπώνουμε σιγά σιγά αυτά τα δικαιώματα, γιατί έχουμε πολλούς εχθρούς Ας πούμε το ISIS δεν έφτασε στη Μοσούλη από τη μία ημέρα στην άλλη. Και γι' αυτό η οργάνωσή μας ασχολήθηκε με αυτό το θέμα μετά από την εισβολή του ISIS. Η οργάνωσή μας, η ε, εκκλησία σε κίνδυνο. Ξέραμε τι συμβαίνει στη Μοσούλη, ήξεραν και οι κάτοικοι, ε, φοβόντουσαν αυτούς τους εισβολείς και δυστυχώς ε, δεν είναι υπέρ της ανεξιθρησκείας. Έχουν και τη δυνατότητα εκφοβισμού. Εμείς θεωρούμε ε, ότι θα σταματήσουν τη δράση τους, αλλά δεν έγινε έτσι. Η ανεξιθρησκεία έχει τρεις διαστάσεις. Το δικαίωμα ύπαρξης ημί θρησκείας, το δικαίωμα ε, αλλαγής θρησκείας και το δικαίωμα να ζει κανείς σύμφωνα με την συνείδησή του ατομικά και συλλογικά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η δήλωση των Ηνωμένων Εθνών αφορά κοινότητες, θεμελιώδη δικαιώματα και μιλάμε για τα δικαιώματα του ατόμου. Τασόμαστε υπέρ αυτής της αρχής στην οργάνωσή μου. Όταν μιλάμε για υπεράσπιση θρησκειών, δεν θα πρέπει να τις εγκαταλείψουμε και να επιβάλλουμε σε ανθρώπους σαν τη Μαρία να ζήσουν όπως θα ήθελε η κοινότητα. Αυτό είναι ακόμα πιο κατασταλτικό γιατί ε, οι, πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι οι αρχές καταστολής έχουν διαφορετικό πρόσωπο, είναι ο εργοδότης σας, η κοινότητά σας. Βλέπετε μία από τις σελίδες εδώ πίσω, μία από τις σελίδες αυτής της εκθέσης, όπως εμφανίζεται στο διαδίκτυο και πρόκειται για αυτό που μιλάμε σήμερα. Υπάρχει ένα παραπέτασμα αδιαφορίας το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτούς που είναι ευάλωτοι, πίσω από τις κοινότητες που ε, στην ουσία βρίσκονται σε κίνδυνο και αγνοούνται τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ε, εκατομμύρια άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Και αυτό το βλέπουμε και, και γύρω ε, στα χίλια χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η πολιτική. Δείτε αυτό τον ε, χάρτη Βλέπετε πώς αναγεννάται ο Άισις σε αυτό το χάρτη. Οι χώρες στο Μαύρο είναι οι χώρες που από το Σεπτέμβριο του 19 οι άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν στην οργάνωση είδαν τις μαύρες σημαίες του ISIS είδαν να δρά το ISIS και να επικρατεί. Και φυσικά με τις ίδιες ομότητες όπως και στο Ιράκ. Ε, είχαμε γύρω στις 4.000 επιθέσεις από ομάδες ε, που βρίσκονται κοντά στο ISIS ή στην Αλκαέδα. Αλκαέντα και στη Μπουρκίνα Φάσο και στη Νιγηρία έδρασαν. Ήρθαν λοιπόν κάτοικοι στους καταβλισμούς μας και στις Φιλιππίνες είναι δραστήριοι όπως σας δείχνω και είναι η υπεύθυνοι για επιθέσεις κατά δύο εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων που έχουν τύχει επιθέσεων και κυρίως βέβαια στρέφονται κατά των ε, γερόντων και των αμάχων, παιδιά και γυναίκες. Στις 15 Φεβρουαρίου, λίγες μέρες πριν, είχαμε την πέμπτη επέτειο του αποκεφαλισμού χριστιανών στη Λιβύη. Η Σύρτη βρίσκεται 850 χιλιόμετρα από τη Βαλέτα από την Λευκοσία στο Ιτλίμπ, γιατί μιλάμε για τις επιθέσεις, η απόσταση είναι 600 χιλιόμετρα μόνο. Κάνουμε λάθος αν θεωρούμε ότι όλα αυτά βρίσκονται μακριά μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ βλέπετε τις χώρες ε, κίτρινο. Πρόκειται για τις ε, αυταρχικές κυβερνήσεις όπου δεν υπάρχει ανεξιθρησκεία. Βλέπε, το βλέπουμε από την Ερυθρέα μέχρι την Ικαράγουα. Όμως η Κίνα με τις δωρεές σε μεγάλα πανεπιστήμια στη Δύση βλέπουμε ότι προωθεί τη δική της πολιτική και καταλαβαίνετε ότι έτσι ε, μας τραβάν το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Θέλετε απλώς να είμαστε παρατηρητές. Η τρίτη πτυχή διακόπτει η ομιλήτρια και λέει κάτι διαφορετικό. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε αυτός ο χάρτης από το Κέντρο Αφρικανικών Σπουδών και είδα ότι αντικατοπτρίζει αυτά που λέμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή πράγματα για τα οποία μας ενημέρωσε η οργάνωσή μας. Γι' αυτό ευεργετούμαστε εάν προβαίνουμε σε ανταλλαγή πληροφοριών εδώ στην Ευρώπη και ξέρω ότι πολλοί ευρωβουλευτές γνωρίζουν την κατάσταση και μπορούμε να σας φέρουμε και μάρτυρες για να σας πούν τι συμβαίνει στην περιοχή τους. Βλέπετε εδώ πώς έχει η κατάσταση γύρω από την Μπουρκίνα Φάσο και την Νιγηρία. Είναι μία πολύ ανησυχητική τάση η οποία θα πρέπει να σταματήσει. Θα θέλαμε να οργανώσουμε μερικά σεμινάρια με στρατιωτικούς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να μιλήσουμε για συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό συνέβη πέντε χρόνια πριν. Αυτό που βλέπετε στην εικόνα. Τι μπορεί να γίνει για να μην ξανασυμβούν τέτοιες δράσεις. Μα τίποτα από ό,τι φαίνεται ε, οι αρχηγοί του ISIS που αποκεφάλισαν τους 21 μάρτυρες από τη Γκάνα και τη Λιβύη δεν θα πρέπει να μπορέσουν να ξαναδράσουν ελεύθερα. Θα ήθελα να σας πω να σας αναφέρω και ένα άλλο θέμα που αφορά την ε, θρησκευτική δουλεία. Μιλάμε για καταναγκαστικούς γάμους αλλά και για εγκλήματα κατά των γυναικών. Αυτά τα εγκλήματα ε, αφορούν και τη Δύση. Μιλάμε για συγκεκριμένες ε, δράσεις κατά των γυναικών οι οποίες αναγκάζονται στη, υποχρεώνονται στη δουλεμπορία οι οποίες απαγάγονται, βιάζονται και μετά μπαίνουν στο κύκλωμα της ε, πορνείας. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες δράσεις και Μιλάμε και για μία τάση γενοκτονίας. Είναι βαριά η λέξη, αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα θέλαμε να αναγνωρίσετε τις συνέπειες αυτών των ε, καταναγκαστικών γάμων και των προσιλητισμών. Ε, λυπάμαι για όλα αυτά τα σκοτεινά σημάδια και γεγονότα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη μάχη αυτή. Η Ευρώπη αρχίζει να αφυπνίζεται και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να ζήσουν σύμφωνα με τις πεπιθήσεις τους. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία της ΕΙΕΔ και τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ θετικά. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη κινείται και υπάρχει και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών με την Εκκλησία, ιδιαίτερα στο Ιράκ και βλέπουμε ότι δυστυχώς η κοινωνία αποδομείται. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η θρησκεία δεν μπορεί να δράσει. Το βλέπετε και στο διαδίκτυο. θεωρώ ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε να δράσουμε πιο ουσιαστικά. Υπάρχει αυτή και αυτή η εξαιρετική έκθεση που φέρει τον τίτλο «Θρησκεία και εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μία εις βάθος ανάλυση». Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να διαβάσετε αυτή την έκθεση και να ε, λάβετε υπόψη αυτή την πραγματικότητα, να ορίσετε έναν πρέσβη ανεξιθρησκείας. Χρειαζόμαστε έναν ειδικό εκπρόσωπο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν πρέσβη καλής θέλησης έτσι ώστε να συνεργαστούμε με όλες τις εκκλησίες και να κατανοήσουμε αυτή την πολυσχηδή διαδικασία. Μετά θα κινηθούμε στην επόμενη, στο επόμενο θέμα, στην επόμενη τραγωδία. Ας λάβουμε υπόψη θέματα συνείδησης και αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Μαρσέλα. Ο κύριος Βαντάλεν. Ο Τζόρτζι, ο Νάτσο, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι καλό το ότι έχουμε αυτήν την ακρόαση για την άνοιξη θρησκεία. Το λέω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα η διαθρησκευτική ομάδα επανασυστήθηκε εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσώπους από όλες σχεδόν τις ομάδες. Οπότε είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Θα ήθελα επίσης να πω πως η κυρία Σιμανσκή ανέφερε κάποια πρακτικά ζητήματα για να μην είμαστε πάρα πολύ ακαδημαϊκοί και έχω το εξής ερώτημα. Πρώτα απ' όλα και στα τρία μέλη του πάνελ. Έχετε μία συμβουλή, μία συμβουλή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι πρέπει να κάνουμε στο θέμα της άνοιξης θρησκείας αν έχετε μία συμβουλή θα μας δώσετε. Το δεύτερο ερώτημα απευθύνεται στον ε, κύριο από την Ιγυρία ο οποίος μίλησε για τοπικό διάλογο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα επιτυχημένου διαθρησκευτικού διαλόγου που έφερε μια αλλαγή στην δική σας τη χώρα αλλά και αλλού που θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα εάν θέλετε για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και άλλα σημεία όπου υπάρχει ένταση μεταξύ των θρησκείων. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Νάτσο. Ε, δεν είναι τόσο ερώτηση όσο σχόλιο. Μιλούμε εδώ για την ε, αναγκαιότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την πίστη του, με την θρησκεία του. Αυτό που φοβούμε είναι μήπως μέσω της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων ε, εισάγουμε εδώ μια θρησκευτική κατεύθυνση, μια θρησκευτική σκέψη στην πολιτική μας ζωή. Γιατί είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη έχει ρίζες χριστιανικές, αλλά ε, το πιο σημαντικό είναι ότι έχει διακρίνει την Εκκλησία από το κράτος ε, και έχει επιτύχει μια κοσμική κατάσταση και εξέταση των πολιτικών της ε, ζητημάτων. Μου φαίνεται λοιπόν ότι να εξετάζουμε κοινωνικά θέματα μέσω της ε, θρησκευτική ε, σκοπιάς είναι θέμα ευαίσθητο. Η κυρία από το Μεξικό αναφέρθηκε στην, στο κορίτσι από, την, από το Τσάπας. Έχουμε παραδοσιακής απόψεις ή αφηγήματα της ζωής και το κορίτσι αυτό ούτε καν σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από γέννημα θρέμα του τσάπας, της περιοχής εκείνης, του τρόπου ζωής. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να διακρίνουμε λίγο την υπεράσπιση των ανθρώπων στα δικαιώματά τους και στις θρησκευτικές τους ε, πεπιθήσεις, χωρίς όμως να επανεισαγάγουμε, επαναλαμβάνω, ε, μία θρησκευτική άποψη της πολιτικής ή της κοινωνικής ζωής, όποια και να είναι η θρησκευτική αυτή ερμηνεία ή δόγμα. Ζητώ να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στη διάκριση των ατομικών δικαιωμάτων της ανεξιθρησκείας, οπουδήποτε στον κόσμο, προσέχοντας όμως πάρα πολύ να μην ξαναλέω εισαγάγουμε μια θρησκευτική απεικόνηση της πραγματικότητας στην πολιτική, στην κοινωνική ζωή. Θυμάμαι και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη χώρα μου που είχε γίνει για την ε, εισαγωγή ε, κάποιων ε, συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και το ζήτημα ήταν δεν μπορούμε να αρνηθούμε το δικαίωμα ενός γονιού να διδάξει τα παιδιά του όπως νομίζει με τις αντιλήψεις του και μπορεί να είναι ρατσιστής αυτός. Αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης τα παιδιά αυτά να γνωρίζουν, να έχουν δυνατότητα να γνωρίζουν ότι έξω από το σπίτι του επικρατούν άλλες απόψεις. Δεν πρέπει δηλαδή να δώσουμε πεδίο ε, υποχώρησης στις ε, κατακτήσεις, στις κοινωνικές ε, και στις ελευθερίες που έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ. και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους. Εγώ είμαι μέλος του Κοινοβουλίου, δεν πρόκειται να σας κάνω μάθημα για τις παραδόσεις του Κοινοβουλίου και τέτοια. Είμαι εδώ για να μαθαίνω από σας και είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για την σημερινή κατάσταση της ελευθερίας πίστης εκτός Ευρώπης ιδιαίτερα. Και πιστεύω, μάλλον μου είπαν οι συνάδελφοι γιατί δεν ήμουν, για την δήλωση του κυρίου ε, Μαχρουντίν Λεμού και τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, ε, γνωρίζουμε όλοι και εσείς και εμείς ότι δεν υπάρχει λύση για όλα, οριζόντια συνολική λύση. Αλλά η θρησκεία είναι γεγονό. Ε, και αλλιώς τη βλέπει κανείς εντός της Ευρώπης και αλλιώς εκτός. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε κάποιες Αντίστοιχε δομές με αυτές που έχουμε στην Ευρώπη, μάλλον δεν ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Ξαναλέω, δεν υπάρχει συνολική λύση. Οι λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν, πρέπει να αναζητηθούν μόνο τοπικά, περιφερειακά. αλλά η θρησκεία και στην Αφρική και αλλού έχει ηθικές τύχες, κοινωνιολογικές πτυχές, έχει έναν παιδαγωγικό ρόλο και πάνω απ' όλα στην διατήρηση της ειρήνης και της επίλυσης κρίσεων, της αποτροπής εντάσεων και συγκρούσεων. Και δεν είναι ότι πρέπει να ελέγξουμε τη θρησκεία καθόλου, πρέπει να τη δούμε ως δυνατότητα. Δεν μιλώ για τη δημιουργία μιας νέας κληρικής τάξης. Ε, το μεγάλο ζήτημα, και ίσως είναι mission impossible, είναι πώς θα το καταφέρουμε. Πώς, τι μπορούμε να κάνουμε ως πολιτικοί, ευρωπαίοι πολιτικοί, επ' αυτού. Θα, με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την άποψή σα σχετικά με τον πιο ενεργή ρόλο που θα μπορούσε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις θρησκευτικέ ελευθερίες. Δεν είναι μόνο θέμα διπλωματίας, να ασκήσουμε πίεση στη ψή, χώρα, τι γίνεται με την τάδε μειονότητα. Μπορεί κάποιο να του ενδιαφέρει αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και δεν είναι προνόμιο ή επικεντρωμένο ενδιαφέρον για τις χριστιανικές μειονότητες που βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Στη Μέση Ανατολή και αλλού, για μένα ως Ευρωπαίος, έχω ιδιαίτερη ευθύνη, αισθάνομαι μια ιδιαίτερη ευθύνη από την παράδοσή μου για τους χριστιανούς. Ε, χωρίς να θέλω να είμαι ακραίος χριστιανός, ταλιμπάν χριστιανός ή κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς υποφέρουν λόγω του απεικιοκρατικού παρελθόντος του ευρωπαϊκού. Υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις χριστιανικές κοινότητες και όταν μιλώ με μουσουλμάνους φίλους, το καταλαβαίνουν απολύτω καλά. Μάλιστα, πολύ συχνά δεν καταλαβαίνουν γιατί τους ξεχνούμε. Πάντως πιστεύω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ο διάλογος. Οι χριστιανικές και μουσουλμανικές κοινότητες όταν συναντιόνται πολύ συχνά λένε απλώς θεωρητικά λόγια τυπικά. Αλλά σε πιο έμπρακτη στήριξη ε, της οικοδόμησης αυτού του διαλόγου. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα η διακήρυξη Αμπου Ντάμπι, ε, το Πανεπιστήμιο Σαλαζάρ, ε, τις δηλώσεις του Πάπα, είναι και αυτές γενικές δηλώσεις, αλλά έχουν τεράστιο αντίκτυπο στους πιστούς. Εμείς ως κοσμικός φορέας, κοσμικό όργανο, πολιτικός φορέας, μπορούμε να λέμε ότι δεν έχουμε σχέση με όλα αυτά, αλλά δεν είναι αλήθεια. Όλα αυτά είναι αποτύπωση της πραγματικότητας. Της πραγματικότητας που υπάρχει μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα που μπορούν να συνοδεύσουν ή να υποστηρίξουν το διάλογο αυτό, το ακαδημαϊκό, το πολιτικό και αυτά θα ήταν πολύ πιο χρήσιμα αντί να κάνουμε διδάγματα το ένα στον άλλο για τις ελευθερίες ε, ανεξιθρησκείας. Ε, άλλες παρεμβάσεις παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους, τα μέλη του πάνελ σας. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις αυτές, πολύ περίπλοκα θέματα. Εγώ θα μιλήσω για τη χώρα που ξέρω πιο καλά, που είναι η Γαλλία. Συμφωνώ απολύτως με αυτή την εικόνα που μας περιγράψατε ε, της γέφυρας μεταξύ των θρησκειών, αλλά πολύ συχνά ε, στη Γαλλία βλέπουμε ότι αυτές οι γέφυρες οικοδομούνται μετά από δυσάρεστες εξελίξεις και πολύ συχνά αποδεικνύονται εύθραυστες. Όταν περνάει η κρίση ή το επεισόδιο, τις ξεχνούμε. Και δεν τις προστατεύει κανείς. Και το είπατε πολύ όμορφα. Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι τι κάνουμε όταν τα πράγματα είναι ήρεμα, γαλήνια, χωρίς ένταση. Ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι όταν έρχεται η κρίση, η ένταση, η αντιπαράθεση. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, πρέπει να μπορούν να συναντώνται οι άνθρωποι και επομένως πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον θα μιλήσουν και χωρίς να έχουμε φόβο ή καχυποψία ο ένα για τον άλλον ή μια ομάδα για την άλλη. Και αυτό που μου έρχεται στο νου στη Γαλλία ε, ε, συζητούσαμε επί τη βάση συγκεκριμένης περίπτωσης ε, το δικαίωμα στη βλασφημία, για παράδειγμα, Εγώ μεγάλωσα σε μια περιοχή που υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορετικότητα και δεν είχαμε πρόβλημα, αλλά σήμερα αυτό που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία δεν επιλύεται τοπικά στη γειτονιά, στην περιοχή, αλλά διαδίδεται μέσω των, του διαδικτύου και παίρνει άλλες διαστάσεις. Τι πιστεύετε εσείς σχετικά με αυτήν την ερμηνεία που ακούμε συχνά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι συχνά δεν μπορούμε ακόμα και ένα ψήφισμα να συμφωνήσουμε ε, προς υπεράσπιση της χι υψή μειονοτικής κοινότητας της θρησκευτική, χωρίς να μας πει κάποιος άλλος ότι ναι, αλλά τότε ξεχνάτε την άλλη κοινότητα και την παράλληλη που είναι πιο μεγάλη και και αυτός ο ανταγωνισμός, αυτός ο τεχνητός κάπως ανταγωνισμός ε, εμποδίζει την προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε γέφυρες. Και λυπάμαι που μακρηγορώ, αλλά με ενδιαφέραν πολύ οι τοποθετήσεις σας. Ε, μιλήσατε και για τον διαθρησκευτικό διάλογο. ε, ε αυτός ο διάλογος αντιμετωπίζει προ, αν θέλετε, προβλήματα αντιπροσώπευσης. Ποιος μιλάει εξ ονόματος κάθε θρησκείας. Τι λύσεις μπορούμε να βρούμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένο δόγμα, αλλά ε, στη χριστιανική εκκλησία έχουμε εκπροσώπους αναγνωρισμένους εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. παρόλα όλα αυτά, ε, πολύ συχνά βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν ταυτίζεται με τους εκπροσώπους αυτούς, τους οποίους όμως αναγνωρίζει το κοσμικό κράτος. Υπάρχει μια εγκατάλειψη η οποία δεν, καθόλου δεν συνεισφέρει στο διάλογο που θα μπορούσε να γίνει. Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο από την Ιγυρία. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση όταν το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο ενέκρινε ψήφισμα για την Ιγυρία, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ αρχής ε, ήθελε να βάλει στο στόχαστρο τους χριστιανούς. Και νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος γιατί τα πρώτα θύματα της Μπόκο είναι οι μουσουλμάνοι και όχι οι χριστιανοί. Και επειδή ομφαλοσκοπούμε ως προς τις χριστιανικές μας ρίζες, φτάνουμε στο σημείο να αρνούμαστε πραγματικά γεγονότα ως προς τα θύματα σε χώρες σαν την Ιγυρία. Νομίζω ότι η προσέγγιση μας στη, στα ε, διαθρησκευτικά ζητήματα στην Ευρώπη δεν ε, γίνεται υπό το σωστότερο πρίσμα. Είπατε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχουν λύσεις χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Έχει μεγάλη σημασία για να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα σας. Η Αφρική ε, ήταν η μία Ήπειρος όπου συνδράμουν όλες οι θρησκείες. Και αυτή η συνύπαρξη ήταν πολύ πιο εύκολη εκεί παρά αλλού. Βλέπουμε όμως ότι γίνεται μια πολιτική, εθνοτική και ε, εθνικιστική μάλλον. Υπάρχει μια ε, εντελώς ε, εθνική, εθνοτική και θρησκευτική προσέγγιση όπου φτάνουμε στο να αρνηθούμε την ύπαρξη μιας θρησκείας. Θα ήθελα να μου πείτε αν κάτι τέτοιο ζείτε σήμερα στην Αφρική και πώς η ιστορία αυτή της συνύπαρξης των θρησκειών σας επιτρέπει να δώσετε απαντήσεις σε αυτή την πολιτική χειραγώγηση που ζείτε και εσείς στη χώρα σας και στην Ήπειρό σας αλλά και εμείς στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Θα αρχίσουμε με εσάς. Έχουμε διερμηνία μέχρι τις 6.30. Ε, ναι. Για την ερώτηση του κυρίου Φαντάλεν για μια συγκεκριμένη συμβουλή αυτό το οποίο κάνουν πολλές ε, χώρες είναι να ορίσουν μια ημέρα ανεξή θρησκείας. Μπορείτε να κάνετε και αυτό εδώ πέρα. Όπως έκανε ο ΙΕ στις 22 Αυγούστου. που λέγεται ημέρα των θυμάτων θρησκευτικής βίας. Αλλά εσείς πείτε το όπως θέλετε. Αλλά καλό είναι να εστιαστεί στην ε, ανεξή θρησκεία. μπορούσε να γίνει όπω γίνεται και στο Κολοσσέο ή στο Κοινοβούλιο Λοιπόν, επίση ε, σημαντικό είναι να καλέσετε εμά ε, για να, προστατε... να προετοιμάσουμε επισκέψει ε, υψηλών αξιωματούχων. Όταν πάτε σε κάποια χώρα να σα ενημερώνουμε εμεί αν όχι εγώ που δεν είμαι στην πρώτη γραμμή, οι συνεργάτε μου που είναι ανά πάση παντού στον κόσμο τώρα. Για αυτό το οποία είπε ο κύριο Σάντσε Αμόρ. θα ήθελα να αναφέρω αυτά τα οποία είπε ο Πατριάρχης ε, Σάκο των Χαλδαίων του Ιράκ που ήρθε εδώ και είπε βοηθήστε μας να αντιληφθεί η Ιρακινή κυβέρνηση ότι πρέπει να διαχωρίσει το κράτος από τη θρησκεία. Μπορείτε να τους πείτε ότι δεν θέλουμε ε, θρησκεία στο κράτος. Αυτό τους βοήθησε να επιζήσουν τελικά. Να διατηρηθεί αυτός ο διαχωρισμός. Ε, είναι θέμα επιβίωσης εκεί. Λοιπόν, αν θέλετε να συνεχίσετε αυτό το επιχειρήμα, οπωσδήποτε στην Μέση Ανατολή θα βρείτε απήχηση, γιατί υποφέρουν ακριβώς επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να διαχωριστεί η Σαρία που τους καθιστά πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Επίσης, να επισημάνω το εξή χτες, ε, η El μια ισπανική εφημερίδα, που δεν θεωρείται φιλική προς την Εκκλησία, υπήρχε άρθρο από την Νιγηρία όπου επέμενε ο δημοσιογράφος για μια πόλη που υφίσταται επιθέσεις από τον μποκοχανόμο ότι φταίει λέει η κυβέρνηση επειδή δολοφόνησε έναν ηγέτη των μουσουλμάνων και μετά ξέσπασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι για χρόνια αισθάνονταν παραμελημένοι από το κράτος. Τότε εδώ πέρα υπήρχε μια θρησκευτική αιτία για την επίθεση του Μπόκο Χαράμ και μας λέει ο άνθρωπος αυτός ότι πριν από 15 μέρες υπήρχε μια επίθεση ε, σταμάτησαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου που πήγαιναν αργά λόγω των λακκουβών που ανέφερε εδώ πέρα ο αγαπητός κύριος. Τους σταμάτησαν λοιπόν από τον Μπόκο Χαράμ, διαχώρισαν τους μουσουλμάνους από τους ε, χριστιανούς 200 χιλιόμετρα αυτό από την πόλη που είπαμε πριν. Άφησαν ελεύθερους τους μουσουλμάνους, πήραν τους χριστιανούς και μετά από λίγες μέρες ε, ανέβασαν ένα βίντεο ε, που τους έβαζαν να γονατίζουν με κόκκινες ε, φόρμες και διάβασαν ένα κομμάτι από το Κοράνι και μετά τους πυροβόλησαν με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Τους χριστιανούς αυτά. Βεβαίω ε, επιθέσει αυτές ξεκίνησαν ε, κατά των εκπροσώπων της ε, κυβέρνησης λόγω της δολοφονίας του ηγέτη τους και μετά επιτέθηκαν κατά στρατού και τώρα στρέφονται κατά των χριστιανών. Σας ευχαριστώ κύριε Μοχαμέτ. Σας ευχαριστώ. Μία σύσταση συμβουλή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν να υπάρχουν πολλαπλά συστήματα εξακρίβωσης δεδομένων. Αν είναι να πιστεύουμε κάτι ως αληθινό, ποτέ να μην ότι ένας δημοσιογράφος είπε «Έχουμε τόσα πολλά fake news στην Νιγηρία, πλασματικά μέσα ενημέρωσης, χρειάζονται πολλαπλές εξακριβώσεις». Έχετε δει στην Ευρώπη θρησκευτικούς πολέμους. Έχετε δει ανθρώπους και χώρες να κάνουν πράγματα στο όνομα του Θεού ή της θρησκείας και γνωρίζετε ότι καμία σχέση με αυτά δεν έχουν. Έχετε εμπειρίες ολοκαυτωμάτων, καταστροφής εκκλησιών από χριστιανούς. Όλα αυτά είναι το να πηγαίνουμε δηλαδή σε μια άλλη χώρα χωρίς να εξετάζουμε προσεκτικά τι συμβαίνει είναι να θυσιάζουμε όλη την πολιτική αυτή παράδοση. Αφενός. Αφετέρου, παραδείγματα επιτυχή διαθρησκευτικού διαλόγου. Εμείς με αριθμό από άλλες οργανώσεις έχουμε συμμετάσχει σε συνεργασίες με θρησκευτικές οργανώσεις που από μια συγκεκριμένη περιοχή επιλέγουν κάποιους θρησκευτικούς ηγέτες, περιοχές που γνωρίζουν ένταση. Το ίδιο κάνουν οι μουσουλμανικές οργανώσεις και μετά τους ε, παρακολουθούν αυτοί οι εκπρόσωποι ε, κάποια προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευση, ενημέρωσης, γιατί πολύ συχνά είναι θερμόεμοι και πολύ συχνά επικρατεί μια αντίληψη στις ομάδες αυτές ότι η θρησκεία μου δεν μου επιτρέπει το α ή το β, δεν μου επιτρέπει να πάω εκεί. Όταν όμως μιλούν μεταξύ τους και κάνουν αυτή την κατάρτιση, δημιουργούν σχέσεις, φιλίες καμιά φορά. Και αυτές οι σχέσεις γίνονται σαν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης. Δηλαδή διαδίδεται το νέο ότι μια εκκλησία καταστράφηκε στη θέση τάδε. Και μετά ρωτάνε τους χριστιανούς ομολόγους τους, είναι αλήθεια και λένε όχι. Και αυτός είναι ένας τρόπος να αποφύγει κανείς την εκδίκηση των, ε, μουσουλ... των χριστιανικών κοινοτήτων που θα ξεσηκώνονταν επειδή καταστράφηκε η εκκλησία ή έτσι κάποιος είπε, διέδωσε. Έχουμε δει τέτοια παραδείγματα σε πολλά μέρη του κόσμου με τέτοια δίκτυα συνεργασίας διαθρησκευτικής. Για το εύθραυστο των σχέσεων αυτών των γεφυρών μεταξύ θρησκειών που είπατε και ότι πολύ συχνά είναι απλώς μια αντίδραση εν θερμό, έχετε δίκιο. Και δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να γίνει φίλος κάποιου άλλου, χρειάζεται χρόνο. Και συχνά σχηματίζουν δεσμούς, σχέσεις. Άλλη φορά είναι όπως αυτό που έλεγα πριν στα το φάρμακο. Δηλαδή χορηγείται αναγκαστικά και τελείωσε. Για, για το ποιος πρέπει να εκπροσωπεί μια θρησκεία. Στον, στην καθολική εκκλησία υπάρχει μια ιεραρχία. Στο, στο, στη σιητική μουσουλμανική θρησκεία επίσης. Στη σουνητική όμως αν στην Ιγυρία, για παράδειγμα, ρωτήσετε ποιος εκπροσωπεί την χριστιανική θρησκεία, τότε θα σας γίνει η διαφημιστική ερώτηση σε ποιο μέρος, για ποιο θέμα. Υπάρχουν ε, εκπρόσωποι, ημάμιδες, υπάρχουν θρησκευτικοί ηγέτες στα διάφορα μέρη. Τα συγκεκριμένα. Στην Ιγυρία αυτό που είπατε για την βλασφημία. Οι σχετικές Διατάξει ή κανόνες που υπάρχουν είναι για να προστατεύουν την ευαισθησία οποιασδήποτε θρησκεία. Δεν είναι μόνο για μουσουλμάνους ή μόνο για χριστιανούς. Για οποιαδήποτε προσβολή κατά του Ιησού, για παράδειγμα, ή του Μωάμεθ, μπορείτε, μπορεί να σας ασκηθεί δίωξη. Αν, αν κανείς θέλει να αστιευτεί, για παράδειγμα, για το τι συνέβη στο Auschwitz, ή τι συνέβη στο ολοκαύτωμα. Κάποιοι θα θεωρήσουν ότι αυτό δεν γίνει επιτρέπεται. Ή αν κάποιο άλλο θέλει να κάνει, ε, να πει ένα ανέκδοτο ε, για, το, για τις 11 Σεπτεμβρίου για την επίθεση στη Νέα Υόρκη. Ε, οι ευαισθησίε υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε και την ελευθερία κάποιου να αναφέρεται σε αυτά. Για την διάκριση κράτους και εκκλησίας αναφερθήκατε αλλά ναι, χωρίς όμως να καταπιέζουμε την Εκκλησία από τους κρατικούς φορείς. Και νομίζω ότι ο, κύριος με κάλυψε σε αυτό. Και πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ποιο κομμάτι της θρησκείας μας φοβίζει όταν αυτό διοχετεύεται στην πολιτική ή κοινωνική συζήτηση. Ας το εντοπίσουμε και ας το αποκλείσουμε αναφερθήκατε και σε κάτι που κάποιοι από εμά παρατηρούμε ως ε, χριστιανική προκατάληψη, δυτική προκατάληψη για τους διωγμούς που υφίστανται μόνο οι χριστιανικές κοινότητες ή ομάδες. Το 90% των θυμάτων της Μπόκο είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή σύμφωνα και με το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Τρομοκρατίας συνολικά τα θύματα είναι 70% μουσουλμάνοι, όλων, όλης της τρομοκρατίας. 90% αυτό, από τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, που έχουν εγκαταλείψει τα χωριά τους, από αυτούς ε, ε, που έχουν σκοτωθεί από την Πόκο Χαράμ, σφαγιαστεί ή που έχουν απαχθεί. Ναι, υπάρχουν παραδείγματα όπως ο αποκεφαλισμός ο ομαδικός που αναφερθήκατε, αλλά έχουμε άπειρα αναρρύθμιτα άλλα παραδείγματα ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την Μπόκο Χαράμ. Οι απαγωγές. Τα κορίτσια εκείνης της περιοχής είχαν και χριστιανές. Είχαν και μουσουλμάνες. Μάλλον υπήρχαν κάποιες χριστιανές, αλλά υπήρχαν δεκάδες χιλιάδων απαγωγές κοριτσιών από μουσουλμανικές κοινότητες που είχαν λάβει χώρα ήδη. Δηλαδή είναι σαν να στέλνει κανείς ένα έμεσο μήνυμα ότι οι μουσουλμάνοι φταίνε για τα όσα συμβαίνουν. Λες και δεν είμαστε και οι δύο κοινότητες θύματα της Μποκοχαράμ. Η Μποκοχαράμ είναι κατά του κράτους. Οποιοδήποτε ε, υπερασπίζεται το κράτο ή το σύνταγμα τη Νιγηρία είναι εχθρό τη. Οπότε σας παρακαλώ, όταν αναφέρετε τα θύματα χριστιανών, αναφέρετε στην ίδια πρόταση και, τα θύματα που ήταν μουσουλμάνοι στο ίδιο επεισόδιο. Δηλαδή, όταν μια ομάδα ένοπλη σκοτώνει τάδε χιλιάδες θύματα χριστιανών, πόσες χιλιάδες μουσουλμάνους έχει σκοτώσει. Γιατί ακούμε πολύ συχνά τέτοιε δηλώσει. Πρέπει να ρωτάμε πάντα πότε, πού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει θρησκευτική προκατάληψη. Υπάρχει στην Ιγυρία όπως υπάρχει και παντού. Αν δείτε πού διαμαρτύρονται ποιε κοινότητε, διαμαρτύρονται εκεί που είναι μειονοτικέ. Στι μουσουλμανικές χώρε διαμαρτύρονται οι χριστιανοί, στις χριστιανικές χώρες διαμαρτύρονται οι μουσουλμάνοι. Και βεβαίως υπάρχουν και εθνικές ομάδες. Υπάρχουν εθνικές ομάδες που έχουν κατοικήσει, επικίσει συγκεκριμένες περιοχές. Και επομένως συνδυάζονται όλα αυτά και με άλλα ζητήματα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε απλά το θρησκευτικό στοιχείο ότι διώκονται επειδή είναι χριστιανοί. Μπορεί να διώκονται επειδή επίκησαν την περιοχή και έρχονταν από αλλού. Για... Ακόμα και στις χώρες που υπάρχει σαρία, νόμος σαρία. Όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ μουσουλμάνου και χριστιανού, ο χριστιανός έχει δικαίωμα να επιλέξει το δικαστήριο στο οποίο θα απευθυνθεί αν έχουμε δύο κλέφτες μουσουλμάνο και χριστιανό ο μουσουλμάνος θα πάει στο δικαστήριο Σαρία και ο χριστιανός θα πάει στο κοσμικό δικαστήριο εκτός και αν υπογράψει ότι συμφωνεί να δικαστεί από δικαστήριο Σαρία. Πρέπει να εξετάζουμε δηλαδή πολύ προσεκτικά ποια είναι τα στοιχεία, τι ακριβώς συμβαίνει για να μην δημιουργούμε εντυπώσει πολιτών δεύτερη κατηγορία, γιατί πάρα πολλοί δυστυχώ έχουν αυτή την εντύπωση. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσα είπαν. Οι συνάδελφοι δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις. Ε, πρέπει να δούμε το τι συμβαίνει επί τόπου. Έτσι θα δούμε το ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί όταν λέμε ότι το θέμα είναι σκεφτικό όταν δεν είναι. Κάποια από αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε, ε, δηλαδή το να περιγράφω κοινότητες με την θρησκευτική του ταυτότητα, ίσως να μην είναι ο καλύτερος τρόπος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Προς τον κύριο Φαντάλεν μια συμβουλή προς το Κοινοβούλιο. Εγώ θα έλεγα το εξής, να συνεχίσετε να στηρίζετε τις πρωτοβουλίες της ε, κυρίας ε, Μογκερίνη και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, αλλά κάντε και κάτι τέτοιο εντός της Ευρώπης. Ο κύριος εδώ σχολίασε τον ρόλο της ε, θρησκείας που είναι πολύ διαφορετικός εντός της Ευρώπης σε σχέση με εκτός στην Ευρωπαϊκή είναι και εντός της Ευρώπης διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο. Οπότε πρέπει να αντιληφθούμε και τις εσωτερικές μας ε, διαφορές και το πώς αυτό διαμορφώνει τον ε, τρόπο με τον οποίο ε, υπάρχει αυτή η διάδραση. Τώρα για τη θρησκεία στη δημόσια σφαίρα. Η διάκριση των εξουσιών ναι, είναι πολύ σημαντική, αλλά το να λέμε ότι η θρησκεία εμποδίζει την πρόοδο νομίζω είναι ένας ε, χοντρικός, μια χοντρική γενίκευση που αγνοεί το πώς ε, η θρησκεία βοήθησε παραδείγματος χάρη να ξεπεραστεί η δουλεία. Αυτό το οποίο εμποδίζει, θεωρώ, την πρόοδο είναι θεσμοί και άτομα που προσπαθούν να δικαιολογήσουν την εξουσία και τα προνομιά τους. Εκεί ε, εμποδίζει η θρησκεία την πρόοδο. Αλλά το ίδιο έχουν κάνει και κοσμικοί θεσμοί. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Όχι το αν κάτι είναι κοσμικό σκεπτικό, αλλά ποιος έχει εξουσία και δεν θέλει να τη χάσει. Για να απαντήσω στα σχόλιά σας ε, σύντομα. Κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι οι δυναμικές της εξουσίας στην παγκόσμια πολιτική και πώς ε, ακούγεται όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάει για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων χριστιανών αλλά όχι για τους μουσουλμάνους στην Κίνα π.χ. ή τη βουδιστική κοινότητα στην Ινδία ή στη Μιανμάρ τη μουσουλμανική κοινότητα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι εικόνα δίνουμε και πώς υπονομεύει την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω λόγο στην εξωτερική υπηρεσία. Um, Εξ ονόματος της ΕΙΕΔ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτή είναι άμεση προτεραιότητα και αυτό που έχει σημασία είναι να ε, δούμε το θέμα της ανεξιθρησκείας που έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μειονοτήτων. Θα πρέπει να μην υπάρχει επίσης υπερβολική, να μην υπάρχουν υπερβολικές κυρώσεις ως προς τη βλασφήμια και πολλές φορές υπάρχουν θρησκευτικά δόγματα τα οποία επιβάλλονται στις ε, μειονότητες, όπως για παράδειγμα η καταναγκαστική γάμη σε μικρή ηλικία. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε σωστές πληροφορίες από ΜΚΟ, ανθρωπιστικές οργανώσεις και να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά μέσα, δηλαδή τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου ε, συζητούμε με τρίτες χώρες σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης ε, θα μπορούσαμε να δούμε θέματα επίθεσης κατά εκκλησιών όπως η ίσχυσε στην περίπτωση της Σρι Λάνκα και του Πακιστάν. Θα πρέπει να ε, αποφύγουμε το ευρωπαϊκό πρίσμα, γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ε, φόρα, τα διεθνή φόρα και τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προωθούμε ένα ψήφισμα και αυτό και με βάση τα δεδομένα του ειδικού η εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών, κάτι το οποίο θα γίνει και τις επερχόμενες εβδομάδες στη Γενέβη. Μέσα στα πλαίσια αυτής της εντολής σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση αυτή. Σας εύχομαι καλό βράδυ εσάβριον.